Κράτη, το σημείο 6, γνωμοδότηση είναι, στις 27 Απριλίου θα εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή για να πάει στο Ιούνιο στο Συμβούλιο και έχει ως εξής το Χρονοδιάγραμμα. Ανταλλαγή απόψεων 22 Φεβρουαρίου. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 26 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Συζήτηση για τις τροπολογίες που έχουν καταδεχθεί στις 16 Μαρτίου. Έγκριση στην Επιτροπή μας 17 Μαρτίου. Έγκριση στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών υποθέσεων 27 Απριλίου. Και Ολομέλεια εκτιμάται στη δεύτερη Ολομέλεια του Μαΐου. Τώρα, το πρώτο θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι η οργάνωση χρόνου εργασίας ε, των εργαζομένων σε οδικές μεταφορές και θα δώσω το λόγο μέσω στην κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα... Πρέπει να σας πω ότι έχω ένα μικρό πρόβλημα, διότι εσείς έχετε λάβει τη τελευταία εκδοχή στη γλώσσα σας πριν από μία ώρα από ό,τι μαθαίνω. Οπότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε το σύνολο τώρα των προτάσεων τροπολογιών που ε, είναι παρακαλώ 100 οι τροπολογίες. Θέλετε να τις συζητήσουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με χαρά να σας πω πώς έχει η κατάσταση. Αλλά επειδή μόλις έχετε πάρει τη μετάφραση. Δεν ξέρω ότι έχει αν έχει μεγάλο νόημα τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειε. Δεν θα αξιολογήσω, ούτε θα κρίνω κάθε πρόταση τροπολογία ξεχωριστά, ούτε θα σα πω ποιε υποστηρίζω και ποιε όχι. Ουσιαστικά αυτό που έχω να σα πω είναι ότι μπορούν να ταξινομηθούν σε τρει ομάδε. Σε τρει κατηγορίε. Την πρώτη ομάδα απλούστατα είναι ή το ένα ή το άλλο οι τροπολογίες. Δεν υπάρχει συμβιβασμός. Στην αρχή, ας πούμε, έχουμε ε, μια σειρά προτάσεων τροπολογιών που ζητούν να απορριφθεί σε λίβδιν η πρόταση. Στη συνέχεια, άλλη ενότητα τροπολογιών, η δεύτερη ομάδα, η κατηγορία, λέγει ότι στην περίπτωση των αυτοαπασχολουμένων, self-employed driver, λέει στα αγγλικά ομιλήτρια, αυτοί θα πρέπει να εξαιρούνται, οι αυτοαπασχολουμένοι. Και αυτή η ε, τροπολογία ε, αποκλεί ε, συμβιβασμό, δηλαδή ή το ένα ή το άλλο εφόσον ζητάει αποκλεισμό. Έχω κάνει και παλαιότερα πρόταση και θέλω να σας πω εδώ ότι έχω να σας προτείνω ξανά κάτι πολύ αξιοπρεπές και πάρα πολύ αποδεκτό. Λοιπόν, οι χώρε εκείνε που θέλουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε να μπουν στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, να είναι ελεύθερε να το πράξουν. Αλλά να μην υποχρεώνουμε κανένα κράτο μέλο να το επιλέξει χωρί να το επιθυμεί. Να μην το επιβάλλουμε, να μην υποχρεώνουμε καμία χώρα να το κάνει. Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ορίζει το χρόνο εργασίας, το ωράριο των αυτοαπασχολουμένων οδηγών. Και νομίζω ότι θα ήταν σφάλμα να ε, προσπαθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξει μέσα από την ομοθεσία αυτή το συγκεκριμένο ωράριο εργασία. Και η τρίτη κατηγορία που σας έλεγα τροπολογιών, ε, μάλλον είναι ε, προϊόν παρεξήγηση ή σφαλμάτων. Γιατί πολλέ τροπολογίε ζητούν να επανέλθουμε στην οδηγία 30 κάθετος 85, οδηγία 30 του 85. Στους συναδέλφους που πρότειναν αυτό στις τροπολογίες τους, έχω να πω το εξής. Και το ζητούν σε διάφορα σημεία του ε, κειμένου και στην τροπολογία 32. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν γίνεται, διότι η οδηγία αυτή έχει καταργηθεί ε, και έχει αντικατασταθεί από την 561. Δεν μπορούμε να έχουμε ως νομική βάση την 30 του 85 διότι δεν ισχύει πια η οδηγία αυτή. Παρακαλώ λοιπόν του συναδέλφου που έκαναν τέτοιε τροπολογίε να τι αποσύρουν. Γιατί είναι σφάλμα, είναι παρεξήγηση, δεν ξέρω, δεν είναι καν αποδεκτέ αυτέ τι τροπολογίε. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία τροπολογιών στις οποίες θα μπορούσαμε ενδεχομένω να βρούμε κάποιο συμβιβασμό, κάποια συνεννόηση και να τις κάνουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Και αυτό θα προσπαθήσω εγώ να κάνω κάθε φορά και εφόσον μπορώ. Στη συνέχεια έχουμε τροπολογίες που είναι αμυγός τεχνικές, με μικρές αλλαγές συντακτικού περιεχομένου και θα προσπαθήσω να τις λάβω υπόψη μου. Σας το υπόσχομαι πραγματικά. Όπου μπορούμε να βρούμε ένα συμβασμό θα προσπαθήσω να τον επιτύχω. Στη συνέχεια τώρα. Υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία από την 104 και επόμενες μέχρι και την τελευταία τροπολογία. Και τι λέγουν αυτές. Εισάγουν νέα μέτρα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο και τα λοιπά, σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για διατάξεις που υπάρχουν ήδη σε άλλα νομοθετικά κείμενα, σε άλλες οδηγίες, σε παραδειγματί. Και ορισμένοι συνάδελφοί που καταθέτουν τις τροπολογίες αυτές, τις ε, δανείζονται από την 561. Υπάρχει όμως και η 1071 που επίσης είναι σχετική και οι συνάδελφοι έχουν βάλει τροπολογίες ε, από την ε, οδηγία αυτή. Θα ήθελα να μάθω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί προς το παρόν αυτά που σας λέω όλα είναι προσωπικές μου απόψεις. Αυτά τα μέτρα δεν ξέρω εάν μπορούν να γίνουν δεκτά υπό όρους και να συστηματοποιηθούν. Δεν είναι προφανές. Αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικές οι τροπολογίες αυτές στη συγκεκριμένη πρόταση. Αφετηρία ποια θα πρέπει να είναι. Ποιος είναι ο στόχος, τι επιδιώκουμε με την πρόταση αυτή οδηγίας. Κυρώσει, παρακολούθηση, έλεγχο. Αυτά που ζητούν λοιπόν οι συνάδελφοι με τις τροπολογίε τους αυτές δεν ε, προκαλούν τίποτα θεωρητικά προβλήματα ή πολιτικά, όχι. Για μένα είναι υπερβολικά τα μέτρα αυτά που προτείνονται. Υπερβολικά αυστηρά, υπερβολικά δρακόντια, αν θέλετε, στην νομοθεσία αυτή. Αντιθέτως, εάν οι περισσότεροι βουλευτές θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά είναι καλά, ότι είναι αναλογικά, ότι δεν το παρακάνουν και ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν ε, διαρριγνύουν την εσωτερική λογική και αρχιτεκτονική του όλου προγράμματος. Ας τις δεχτούμε και στην τελευταία, στην τελική ψηφοφορία θα δούμε τι θα γίνει. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα. η οριστική ψηφοφορία προβλέπεται να γίνει στη δεύτερη ολομέλεια του Μαΐου. Θα παρακαλούσα, και το έχω ήδη ζητήσει από τη γραμματεία, θα παρακαλούσα, λέω, να προσαρμόσουμε έτσι το χρονοδιάγραμμά μας και τις συζητήσεις ε, γύρω από αυτή την πρόταση. Γιατί το λέω αυτό. Ουσιαστικά μία εβδομάδα μας μένει για να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Στις 4 Μαρτίου θα πρέπει να ψηφίσουμε εμείς και η οριστική ψηφοφορία στην Επιτροπή μετά από δύο μήνες. Γι' αυτό λέω τις συμβαστικές τροπολογίες να μην τις συζητήσουμε στις 4 του μηνός αλλά στις 16 και μετά θα έχουμε αρκετό χρόνο στις 25 Απριλίου να το ψηφίσουμε. για να γίνουν και οι ε, μεταφράσεις μέχρι τη δεύτερη ονομέλεια του Μαΐου. Αυτά εισαγωγικά, Πρόεδρε, και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ. Έχω έναν ομιλητή, τον κύριο Κλάρκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ήδη γνωρίζουμε και εκτιμούμε ότι οι αυτοπασχολούμενοι οδηγοί θα πρέπει να συμμορφούνται προς τις υπόλοιπες γενικές οδηγίες ε, όσον αφορά το χρόνο οδήγησης. Ε, αυτό που μας ανησυχεί είναι τι κάνει ο οδηγός στο χρόνο του ως αυτοπασχολούμενος οδηγός, όπου αναμφίβολα εργάζεται σπίτι του με έναν υπολογιστή ή άλλους ε, πόρους, εργάζεται, φτιάχνει νέο χρονοδιάγραμμα, βρίσκει νέους πελάτες και, εν πάση περιπτώσει, διασφαλίζει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί. Και είναι όπω και εμεί εδώ οι ευρωβουλευτέ. Πάμε σπίτι μα και κάνουμε και εκεί δουλειά. Δεν μιλάω στο γραφείο μα, μιλώ για το σπίτι μα. Ποιο μα παρακολουθεί για το τι κάνουμε. Δεν είναι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τους αυτοαπασχολούμενου οδηγού στο σπίτι του που κάνουν ό,τι χρειάζεται να κάνουν ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τη δουλειά του, ώστε να διατηρήσουν δηλαδή την απασχόλησή του. Και είμαι βέβαιο ότι όλοι συμφωνούμε πω θέλουμε να διατηρήσουν την απασχόλησή του και δεν θέλουμε να ε, βρεθούν ε, άνεργοι, ούτε θέλουμε να τους οδηγήσουμε στις αγκάλες των μεγάλων ε, ομίλων και να τους κάνουμε απασχολούμενους ή μάλλον υπαλλήλου. Θέλουμε να έχουμε αυτοαπασχολούμενους οδηγούς που είναι άνθρωποι που εργάζονται για τον εαυτό τους στον κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους επίσης. Συμφωνεί μαζί μου φαντάζομαι και η η συγχύτρια και γι' αυτό και προτείνω στην Επιτροπή να, να απορρίψουμε αυτή την οδηγία όπου και να επανέλθουμε στην αρχική όπου ούτως ή άλλως οι αυτοποσχολούμενοι εξαιρώνται. Ευχαριστώ κύριο Σέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάουερ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι σχέση, σε σχέση με τις πρωτοβουλίες σας, μάλλον την πρόταση, να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες εξ ονόματος της ομάδας μου. Εάν δεν διαφωνούν οι διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής, δεν μας φαίνεται κακή ιδέα, γιατί όχι, 16 Μαρτίου, για να ψηφίσουμε στις 25 Απριλίου. Γιατί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η οδηγία αυτή θα πρέπει να κανονιστεί, να συζητηθεί ε, κατά τη διάρκεια της συνεννόησης για τις συμβιστικές τροπολογίες μεταξύ της εισηγήτριας και τους σκιώδη εισηγητές. Αν δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, συμφωνώ να, ναι, να μην μπούμε σήμερα ε, στις 100 τροπολογίες στην ουσία τους, γιατί τα επιχειρήματα τα ξέρουμε πάρα πολύ. Αυτό μου θυμίζει το ψυχρό πόλεμο, κύρια Μπάουερ. Οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι κάνανε ε, συνέχεια τα ίδια επιχειρήματα, έλεγαν οι Ρώσοι. Επιχείρημα 1. Οι Αμερικανοί απαντούσαν ωραία. Απάντηση νούμερο 2. Πάμε στο επόμενο. Και έτσι πήγαινε η ιστορία με τα νούμερα και δεν χρειαζόταν καν συζήτηση. Ξέρανε και το ερώτηση και την απάντηση από τα νούμερα. Και ε, τα ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς πιστεύουμε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να παραμένουν στην οδηγία. Και το αντιπεχείρημα πάντα ήταν ότι «Αμα είναι πολύ δύσκολο να τους ελέγξεις». Όπως είπε ο κύριος Κλάρκ τώρα, κάνουν και άλλη δουλειά εκτός ε, τιμονιού, εν πάση περιπτώσει, και, και εκτός ε, του πεδίου της οδηγίας. Δεν είναι θέμα ούτε κόπωσης, ούτε τροχαίων, γιατί δουλεύουν και στο σπίτι τους. Παρακαλώ κύριε Μπάουρ, κοιτάξτε ε, τις ε, τροπολογίες των σοσιαλιστών ε, όπου ζητούμε διευκρίνηση. Να πούμε ε, ξεκάθαρα ότι μιλούμε ακριβώς μόνο για τους χρόνους οδήγησης, μόνο για αυτό μιλάμε και ε, μόνο για σωματική εργασία φορτοεκφόρτωσης. Αυτό που σημαίνει σωματική κόπωση, δηλαδή άρα και κίνδυνο για την ασφάλειά του και για την ακεραιότητα των οδηγών στον αυτοκινητόδρομο. Ξέρουμε τα επιχειρήματα, επανειλημμένα τα έχουμε ακούσει, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι είναι στο, αν είναι στο πεδίο της εφαρμογής της οδηγίας αυτή σημαίνει άπειρη γραφειοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι αν κοιτάξετε τις δικές μας τροπολογίες ακριβώς προσπαθούμε να ελέγξουμε αυτό που ελέγχεται μόνο από τον ταχογράφο. Ε, με μια μικρή ίσως αναφορά σε μια καταποκοπή ε, μορφή ελέγχου, ε, άπαξ εβδομαδιαίας ας πούμε, αλλά υπάρχουν και ψευδό αυτοαπασχολούμενοι και τα ξέρουμε. Και το ίδιο πρόβλημα ελέγχου είναι και η ίδια δυσκολία. Αν είναι δύσκολο να ελέγξεις πόσο εργάζεται ένας αυτοαπασχολούμενος, εξίσου δύσκολο είναι για τον ψεύδο απασχολούμενο που εμφανίζεται ως υπάλληλο. Ή που είναι υπάλληλο και εμφανίζεται ως απασχολούμενος μάλλον ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα τροχιά, τους κινδύνους ε, στον αυτοκινητόδρομο. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ύπαρξη συνθήκων εργασίας με στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μας και των εταιριών μας. Να βάλουμε παντού κανόνες για να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ εταιριών. Για τη δεύτερη ενότητα τροπολογιών τώρα θα ήθελα να σας πω το εξή. Είναι γεγονός ότι θα μπορούσε μία διέξοδος εδώ να είναι να αφήσουμε ελεύθερο κάθε κράτος μέλος. Και αυτό θα μας έλυνε μερικά προβλήματα. Να αποφασίζει το κάθε κράτος μέλος κατά πόσο οι αυτοαπασχολούμενοι εντάσσονται ή όχι στην οδηγία. Θα σας παρακαλούσα όμως να σκεφτείτε το εξής κυρία Μπάουερ. Αυτό λύνει ένα μέρος μόνο του προβλήματος. Αλλά οι αυτοπασχολούμενοι δεν εργάζονται μόνο σε ένα κράτος, διασχίζουν σύνορα. Οπότε λογικό δεν είναι να πούμε ότι είναι εθνικό το ζήτημα. Ε, μάλλον δεν είναι μόνο εθνικό αλλά ευρωπαϊκό. Αν ένας Ισπανός κουρασμένος οδηγός οδηγεί στη Γαλλία, δεν είναι λογικό να απαιτούμε ε, οι κανόνες που τον διέπουν να είναι οι γαλλικοί κανόνες και όχι κάθε χώρα να έχει κατά το δοκούν ό,τι θεωρεί σκόπιμο. Είναι πολύ σημαντικά θέματα η ασφάλεια στον αυτοκινητόδρομο και η υγεία. Δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση εδώ βάσει της εθνικότητας. Γιατί έτσι είναι ακόμα ε, πιο δύσκολος ο έλεγχος. Θα πρέπει η τροχέα να ξέρει την νομοθεσία 27 κρατών μελών. Για να δω τι είσαι εσύ που σε σταματάω να σε ελέγξω. Τσέχος, Σλοβάκος, Ούγγρος, Ρουμάνος, Φιλαδός και πάει λέγοντας. Δεν είναι λύση αυτή. Ό,τι και να κάνουμε τελικά στο ίδιο πρόβλημα προσκρούμε. Και το πρόβλημα είναι ότι αν έχουν όλοι τον ίδιο κανόνα ή αν θεωρήσουμε ότι μπορούν να έχουμε διαφορετικούς κανόνες για να οδηγούμε στους αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη. Οπότε, κυρία Μπάουε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τα εξή πράγματα και πολλά. Πρώτον, να συζητήσουμε αυτό, ότι χωράει η συζήτηση, εφόσον θα έχουμε λύσει το θέμα της ουσίας που είναι οι τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στην απόσυρση από την οδηγία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολουμένων, όπως έχει τώρα. Κυρία Πρόεδρε, εμεί είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε κάθε λογικό συμβιβασμό που θα χρειαστεί αν χάσουμε επί της ουσίας αυτό που ζητούμε. Αλλά είναι πιο λογικό να ορίσουμε καλύτερα τι εστί αυτοπασχολούμενος, για να μην υπάρχει κατάχρηση αυτής της μορφής εργασίας. Για να... Ε, κάναμε λοιπόν τροπολογίες για να είναι η έλεγχη πιο αποτελεσματική, ποιος είναι αυτοπασχολούμενος, ποιος είναι υπάλληλο και να παρακολουθείτε σωστά η οδηγία να βλέπουμε, να διδασκόμαστε και από τις επιτυχίες και από τις αποτυχίες μας. Εμείς διατηρούμε τη θέση μας επί της αρχής. Αν λυθεί όμως αυτό και αν δεν πετύχουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι και κοινή λογική και νομική λογική, θα μπούμε και στη συζήτηση για τις συμβαστικές και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να το συζητήσουμε με την εισηγήτρια. Και στην Α και στη Β υπόθεση αυτό που μας ενδιαφέρει στην Ευρώπη να είναι καλύτερη η οδηγία και η καλύτερη κατάσταση από τη σημερινή. Ευχαριστώ πολύ. Um, uh, σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκέψη πίσω από την οδηγία αυτή είναι να βελτιώσουμε την ασφάλεια στους δρόμους μας. Μια και σκεφτόμαστε την οδική ασφάλεια, το βασικό ερώτημα είναι οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με τα ωράρια οδήγησης. Θα πρέπει να γίνεται ε, καλή επιτήρηση και αυτή αναπόκειται στα κράτη-μέλη. Είναι σκανδαλώδες το ότι δεν έχουμε βάση δεδομένων, δεν έχουμε κάποιο ε, έλεγχο των πληροφοριών σε διασυνοριακό επίπεδο. Και ισχύει αυτό που υπόθηκε, ότι ένας οδηγός μπορεί μέσα στο ίδιο 24ωρο να περάσει από πολλά κράτη-μέλη και να τον ελέγξουν αρκετές, διάφορες αρχές, οι αρχές διαφορετικών κρατών μελών. Φυσικά η οδήγηση ε, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας στα πλαίσια της ε, οδηγίας αυτής έχει συζητηθεί και ότι η φόρτωση και εκφόρτωση ε, είναι σημαντικό θέμα και επηρεάζει πολύ την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Ε, θα θέλαμε να ξέρουμε τι πιστεύει η Κομισιόν, πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε τον ε, χρόνο οδήγησης. Θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιες λεπτομέρειες αναλυτικά, διότι είναι σαφώς ότι ε, στόχος ε, όλων των οδηγιών είναι να λύσουν προβλήματα, όχι να δημιουργήσουν προβλήματα και θα πρέπει να θέσουμε το εξή ερώτημα. Οι ανεξάρτητοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε θα πρέπει να εμπίπτουν στην οδηγία ή όχι. Και είναι σημαντικό το τι απαντήσει δίνει η οδηγία αυτή στα ερωτήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των διαβολεύσεών μα. Ε, άλλο θέμα που προκύπτει είναι οι δίθεν, ε, ανεξάρτητοι, ε, οι δίθεν ελεύθεροι επαγγελματίες στην ε, χώρα μου, στην Φιλανδία, δεν είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Ξέρω όμως ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι σοβαρό το πρόβλημα. Στην οδηγία αυτή λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η σκέψη ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερο έλεγχο και θα πρέπει να σφίξουμε τα κριτήρια, να τα κάνουμε πιο αυστηρά. Άλλοι συνάδελφοι έχουν υποβάλει προτάσεις ε, ε, σχετικά με το ότι ο, ελεύθερος, ο ανεξάρτητος επαγγελματίας δεν ε, θα πρέπει να εξαρτάται οικονομικά από κάποιον άλλον. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, διασφαλίζουν τον εντοπισμό των ε, σωστών ελεύθερων επαγγελματιών. Είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια οδηγία που θα μας επιτρέψει να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Eh, Ευχαριστώ, κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Ε, νομίζω ότι είναι βαρύ το έργο που έχει μπροστά της. Πιστεύω όμως ότι θα πετύχει ένα συμβασμό που θα αξίζει τον κόπο. Ε, κάποιες παρατηρήσεις. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Σέρκας, δεν χρειάζεται να, να επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα. Έχουν ε, αναφερθεί επανειλημμένα. Όσον αφορά τις ε, προτάσεις τροπολογιών για την καταπολέμηση του προβλήματος των Δήθεν... Ε, ανεξάρτητων επαγγελματιών. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια και όπως είπε είναι πρόβλημα το οποίο ε, δεσπόζει σε κάποια κρατημέλη, όχι όμως σε άλλα. Ε, εγώ θα ήμουν διατεθειμένη να προωθήσω κυρώσεις ή ό,τι είναι απαραίτητο για να πετύχουμε κάποιον συμβιβασμό ένα θέμα που δεν αναφέρθηκε, ε, το, για το οποίο όμως έχουν υποβληθεί σχετικές τροπολογίες, είναι η συμπερίληψη των ε, οχημάτων ε, κάτω των 3,5 τόνων η συγγήτρια είπε ότι αν ε, αυτό ε, δικαιολογείται από κάποια μελέτη σκοπιμότητας, τότε θα μπορούσε να γίνει αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν σχετική μελέτη επιπτώσεων, μελέτη σκοπιμότητας. Ε, και επίσης όσον αφορά τους ταχογράφους, θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα αυτό. Το να αφήσουμε στα κράτη-μέλη την τελευταία κουβέντα δεν θα είναι εύκολο δεδομένου του ανταγωνισμού, δεδομένου των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Και κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις. Ε, θα πρέπει στην ε, συζήτηση αυτή να θυμόμαστε ότι έχουμε τους ίδιους κανόνες για χρόνο οδήγησης και χρόνο ανάπαυσης σε όλα τα κρατημέλη Και η τελευταία μου παρατήρηση. Κάποιες τροπολογίες, για παράδειγμα η 89 και κάποιες άλλες αναφέρονται στη συμπερίληψη νέου σημείου στο άρθρο 4. Λένε ότι ε, ο χρόνος που αναφέρεται στο άρθρο 3 3-2, ε, που αναφέρεται στις δραστηριότητες 3, 4 και 5, θα πρέπει να είναι μία ώρα τη βδομάδα, άλλοι είπαν δύο ώρες τη βδομάδα. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούμε εδώ. Λέμε ότι αν αποφασίσουμε τώρα σε κάποια χρονική περίοδο αυτό θα είναι άσχετα από το αν ο κόσμος ε, τελικά δαπανεί 6 ώρες ή 10 ώρες ή μισή ώρα. Δηλαδή θα θεωρείτε ότι ο χρόνος ε, εργασίας είναι ε, μία ώρα επειδή το λέμε εμείς. Εμένα μου φαίνεται περίεργη η τροπολογία αυτή διότι είτε η αιτιολόγησή μας είναι η κούραση οπότε δεν μπορούμε να θέσουμε όριο διότι μπορεί κάποιος να χρειάζεται 10 ώρες και όχι μία. Και αν αυτή είναι η πραγματική μας ανησυχία, τότε δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες που να ορίζουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο να μην έχει καμία σχέση με το πραγματικό χρονικό διάστημα που απαιτείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντέλη. Ε, euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος συναδέλφου Εμιλή Τουρινέν που είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη θέση της ομάδας των Πρασίνων. Στα αγγλικά θα σας τα πω. Αποφασίσαμε να επανυποβάλλουμε την πρόταση για απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν γιατί θεωρούμε πως η συμφωνία στην οποία έχει φτάσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι χρήσιμη για τον τομέα των μεταφορών ώστε να διασφαλιστεί η θυμητός ανταγωνισμός. Το 2002 συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί μέχρι τις 23 Μαρτίου 2009 και σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου οι αυτοαπασχολούμενοι συμπεριλαμβάνονται τώρα και τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουν εφαρμόσει τα σχετικά μέτρα. Μόνο δύο χώρες όμως το έχουν κάνει αυτό. Αυτό το σαφές μήνυμα από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου υπογραμμίζει μια προοπτική. Εδώ δεν μιλάμε για την συμπερίληψη των αυτοπασχολούμενων, γιατί ήδη συμπεριλαμβάνονται και δι' από την οδηγία. Μιλάμε για την εξαίρεση αυτών. Αυτή η κατάσταση, αυτή η νομική διαδικασία και αυτή η διεθνής θεσμική ε, ιστερία στην ορχησία δείχνει μια κομισιόν που απλά δεν σέβεται το κοινοβούλιο και την απόφαση που έχει λάβει. Πρόκειται για ένα σοβαρό δημοκρατικό πρόβλημα. Δεν είμαστε κοινοβούλιο που θέλει την επανυποβολή ε, της οδηγίας κάθε φορά που δεν Πακούμε ε, στις δικές της υποδείξεις. Όμως, διακυβεύονται πολλά περισσότερα για τους ίδιους τους οδηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εργάζονται σε έναν ελεύθερο τομέα με ένα σωρά προβλήματα όσον αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, το χρόνο οδηγηση, την παρακολούθηση αυτού. Οι οδηγοί είναι αυτοί που θα έπρεπε να μας απασχολούν αυτή τη στιγμή και στους οποίους θα έπρεπε να ενδιαφερόμαστε. Έχουμε υποβάλει την τροπολογία 17 για την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν. Ίσως να μην έχουμε πλειοψηφία, αλλά ξέρουμε πως πολλοί κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν δεν είμαστε πλειοψηφία, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στις δυνατότητες συμβιβασμού, αλλά δεν μπορούμε σε, κάθε περίπτωση, σε καμία περίπτωση να συστήσουμε την αποδοχή αυτής της οδηγίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μπω σε μερικά σημεία της προλαλής σας. Και ε, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα που λέει που να ξέρει η αστυνομία τι ισχύει σε ποια νομοθεσία, σε ποια χώρα. Αυτό παντού υπάρχει στην Ευρώπη δεν χρειάζεται κάθε αστυνομία να γνωρίζει τι γίνεται στην άλλη χώρα. Τι θα κάνουμε, είτε θα κατεβάσουμε ρολά στην Ευρώπη, είτε ε, θα γίνουμε ένα κράτος όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε αυτό το θέλουμε. Αυτό το επιχείρημα λοιπόν λίγο με προβληματίζει εμένα και με δυσκολεύει. Ε, παρακαλώ να δείξετε λίγη κατανόηση για τη συζήτηση που κάνουμε για τους ψευδοαυτοαπασχολούμενους. Ε, έχουμε ε, ορισμένους που ήδη εργάζονται έτσι με αυτό το καθεστώς και κάποιους άλλους που αναγκάζονται και εξωθούνται προς την αυτοπασχόληση, την ψευδή. Έχω κάνει μια τροπολογία με αριθμό 28 και σας τη συνιστώ και ως ε, συμβιβαστική και λέει ότι οι μεταφορείς θα πρέπει να παραμείνουν εκτός του συστήματος. Ο επιχειρηματίας ο ίδιος, ο οποίος έτσι και υφίσταται ε, και διέπεται από την οδηγία αυτή να παραμένει, αλλά αν αλλάξει τίποτα, να αλλάξει και η νομοθεσία, αν αλλάξει κάτι στο καθεστώς, Για να προχωρήσουμε λίγο ε, με αυτή την υπόθεση των ψευδός αυτοαπασχολουμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Βέκνερ. Heute in der Nacht. Äh, χτες το βράδυ στο εξωτερικό δακτύλιο της ε, ε, Βιέννης έγινε ένα δυστύχημα με ένα λεωφορείο και δύο φορτηγά. Αποτέλεσμα 6 νεκροί και 37 τραυματίες. Νύχτα έγινε το όλο και διαπιστώνει η αστυνομία ότι πρόκειται για ένα δυστύχημα γιατί αποκοιμήθηκε ένας από τους οδηγούς του φορτηγού για δευτερόλεπτα. Δηλαδή ε, ε, δευτερόλεπτα σε παίρνει ο ύπνος και έχεις 6 νεκρούς και 37 τραυματίες. Ακούγονται διάφορα επιχειρήματα ε, ε, και εξαντλητικά μάλιστα περιγράφονται, αλλά βλέπουμε το παράδειγμα αυτό πόσο θλιβερό είναι και πόσο ε, στους κανόνες αυτούς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι, γιατί η ασφάλεια και η ακαιρεότητα όλων των επιβατών ε, και η των ίδιων των οδηγών φορτηγών θα πρέπει να διασφαλίζεται και να παραμένει ε, στο επίκεντρο. Και η οδηγία 15 του 2002 είναι ε, εφαρμοστέα ένα χρόνο μόνο. Δεν έχουμε ε, πολλά στοιχεία για να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη και ποιες είναι οι συνέπειες και οι επιπτώσεις στην ασφάλεια και στην ακαιρεότητα ε, όλων των ενεχομένων στην κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους. Θα πρέπει να γίνει μια μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα. Ήδη από τώρα δηλαδή να θέλουμε να βάλουμε τους αυτοπασχολουμένους στην οδηγία δεν ε, είναι σκόπιμο ούτε από πλευράς χρονικής ούτε γενικότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Μπάουερ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν απευθείας προς εκείνη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ας είμαστε σαφείς η ασφάλεια στους δρόμους αλλά και η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι κύριο μέλημα της Κομισιόν και διέπει όλες τις προτάσεις που κάνει. Εδώ όμως δεν μιλάμε περί αυτού. Μιλάμε βασικά για την αποφυγή του κινδύνου των αυτοαπασχολούμενων οδηγών ε, να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ε, από πλευράς των ε, εργοδοτών τους. Έχω ήδη μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής αρκετές φορές και όπως είπε και ο κύριος Σέρκας, έχουμε ανταλλάξει επιχειρήματα τόσο συχνά που δεν έχει νόημα να επανερχόμαστε και να επαναλαμβανόμαστε. Γι' αυτό θα εστιάσω την προσοχή μόνο στις τροπολογίες και... Αν παρόδο θα απαντήσω και στις ερωτήσεις που ετέθησαν πρώτον. Όπως είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, η Κομισιόν υποστηρίζει τις, τις ε, τροπολογίες της κυρίας Μπάουερ και θεωρεί ότι οι τροπολογίες που έχει υποβάλει θα είναι πολύ χρήσιμες για την αποσαφήνιση ενός κειμένου που ίσως να δίνει λαβή σε διαφορετικές ερμηνείες και διαφορετική μεταχείριση στα διάφορα κράτη-μέλη. Οι τροπολογίες της κυρίας Μπάουερ λοιπόν υποστηρίζονται όλες από την Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες που κατά την άποψή μας επιβάλλουν δυσανάλογο διοικητικό φόρτο και κόστος στους επιχειρηματίες και στα κράτη-μέλη. Ενώ δεν προβλέπουν επαρκή μέσα ελέγχου εφαρμογή της οδηγίας, της ε, νομοθεσίας όσον αφορά τους πραγματικά αυτοπασχολούμενους οδηγούς που συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Είμαστε αντίθετοι προ αυτέ τι οδηγίε, αν και αναγνωρίζουμε ότι ο Χιούς και ο κύριος Ελκαντράουι που είναι εισηγητής για την γνωμοδότηση στην Επιτροπή Μεταφορών έχουν καταβάλει προσπάθεια για εξέβρεση συμβιβαστική λύσης όσον αφορά τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών αλλά ίσως με ένα ε, καταποκοπήν όριο μιας δυο-τριών ωρών για την ε, εργασία γραφείου ας πούμε. Αυτή είναι η συμβολή του στην οδηγία για το χρόνο απασχόλησης. Ωστόσο οι τροπολογίες αυτές όποια και αν πρόθεσή τους δεν λύνουν το θέμα της ε, επιβολής και της εφαρμογής της ε, νομοθεσίας. Γιατί όπως σας έχω ήδη εξηγήσει, το μόνος τρόπος που έχουμε αυτή τη στιγμή για να επιβάλλουμε επιπλέον χρόνο εργασίας, επιπλέον του χρόνου οδήγησης, είναι ο ταχογράφος. Και όταν ε, και ενώ οι υπάλληλοι οδηγοί έχουν συμφέρον να χρησιμοποιούν τον ταχογράφο όταν φορτώνουν εξελτώνουν το φορτηγό και δεν οδηγούν ή αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν τέτοιο συμφέρον και κίνητρο. Και άρα, εκτός και αν δημιουργήσουμε φοβούμε ένα πολύ ε, βαρύ σύστημα ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα είμαστε σε θέση να... Μάλλον τα κράτη-μέλη δεν θα είναι σε θέση να ελέγξουν εργασία εκτός της οδήγησης για τους αυτοπασχολούμενους. Άρα λοιπόν οι τροπολογίες που αυτό το στόχο έχουν είτε για τη συμπερίληψη είτε τη συμπερίληψη αλλαγών με επιπλέον ε, μορφές ελέγχου είναι τροπολογίες που δεν μπορούμε να στηρίξουμε ως Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετές τροπολογίες όπου η Κομισιόν τη στηρίζει και προέρχονται από διάφορες πολιτικές ομάδες. 20 με 23, 28, 29, 31, 33 με 36, 38, 40 με 48, 54, 56, 60, 68, 71, 76, 97. Όλες αυτές είναι τροπολογίες που βελτιώνουν τη σαφήνεια των διατάξεων και βελτιώνουν τη δυνατότητα επιβολής του νόμου. Ανάμεσα σε αυτές τις τροπολογίες υπάρχει και μία που αφορά τους 3,5 τόνους και το σχετικό όριο. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά όπως έχω ήδη πει, νομίζω πως θα πρέπει να ε, το εξετάσουμε γενικότερα. Δηλαδή, στην νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διάφορες νομοθεσίες, κανονισμοί, οδηγίες και που όλοι ε, ισχύουν για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Και αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Κάτω από αυτό δεν καλύπτεσαι, πάνω από αυτό καλύπτεσαι. Αν, αφήσουμε, αν αλλάξουμε λοιπόν το όριο των 3,5 τόνων, μπορούμε να το πράξουμε μόνο αν το κάνουμε γενικώ και με συνέπεια. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτή την ιδέα, τη μελετούμε μάλιστα και γίνεται αυτή τη στιγμή μια έρευνα, μια μελέτη και κάνουμε ένα σωρό μελέτες αξιολόγησης και αντίκτυπου κτλ. Και αν δούμε τελικά πως υπάρχει νόημα στο να διευρύνουμε το όριο να το μειώσουμε δηλαδή κάτω από τους 3,5 τόνους, θα κάνουμε και τις αντίστοιχες προτάσεις. Να πω ακόμα δύο λόγια για τις τροπολογίες 35 και 36 που έχουν κατατεθεί από την κυρία Γιά Κονσάρη. Είναι ενδιαφέρουσες και θα τις μελετήσουμε πιο ενδελεχώς. Η 35 προτείνει το να θεωρηθούν υπεύθυνοι οι αυτοπασχολούμενοι οδηγοί για τις υπερορίες που κάνουν αν αυτό αποδειχθεί πως έχει οδηγήσει σε κίνδυνο. Στη 36 λέει κάτι το οποίο σχολιάστηκε ήδη, ότι δηλαδή τη δυνατότητα αυτομάτως να θεωρήσουμε εργασία που δεν είναι δουλειά στο τιμόνι, δεν είναι οδήγηση, που είναι φόρτωμα, ξεφόρτωμα του φορτηγού. Όπως είπα, ήδη τώρα υπάρχει νομικά η υποχρέωση να καταγράφονται αυτές τις δραστηριότητες ως άλλη εργασία. Όμως εξαρτάται από τον συγκεκριμένο οδηγό και τον αυτοαπασχολούμενο να πατήσει το κουμπί. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πώς θα είμαστε βέβαιοι πως τα κράτη-μέλη θα επιβάλλουν μια τέτοια νομοθεσία που ήδη υπάρχει. αυτόματη καταγραφή των δραστηριοτήτων φορτωση εκφόρτωσης θα έλυνε το πρόβλημα της ακρίβειας καταγραφής των ορών εργασίας, αλλά πρέπει επίσης να σημειώσετε ότι η φόρτωση εκφόρτωση είναι κάτι που εξαρτάται πολύ από τα συγκεκριμένα φορτία ε, και δεν ε, εξαρτάται από τον οδηγό τον υπάλληλο ή τον αυτοπασχολούμενο, δεν είναι πάντα ο ίδιος που φορτώνει ή ξεφορτώνει, οπότε επανερχόμαστε σε ένα πολύ περίπλοκο θέμα επιβολής υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να καλύψει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή οποιαδήποτε νομοθεσία, αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Μπάουερ για να κλείσουμε τη συζήτηση, να πω ότι η Γραμματεία εξέτασε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και είναι δυνατόν να συζητήσουμε τις συμβιβαστικές στις 16 Μαρτίου και 28 Απριλίου να κάνουμε την τελική συζήτηση. Υπάρχουν ίσως κάποια μικρά προβλήματα. Αν υπάρξουν θα σας ενημερώσουμε. Κυρία Μπάουερ, έχετε το λόγο για να συνοψίσετε. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που προσπάθησαν να βελτιώσουν την έκθεση. και που δαπάνησαν χρόνο για την έκθεση αυτή. Εκτιμώ τις προσπάθειές τους, καθότι αρκετοί συνάδελφοι έκαναν σαφή τη θέση τους. Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Ε, ο κύριος Στέρκας είπε ότι Σέρκα είπε ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά με το επί θέμα και μετά μπορούμε να συμφωνήσουμε για όλα τα άλλα. Θα ε, ευχαριστούσε πολύ αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Νομίζω όμως ότι αυτό ε, θα γίνει σαφές ε, στο τέλος. Δυστυχώς, όπως όλοι ξέρουμε, μπορεί να μην Ε, γίνει αυτό τελικά. Το πρόβλημα με τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων είναι ένα θέμα το οποίο ε, έχει τεθεί και στη δική μας Επιτροπή και στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, καθότι ε, έχει αλλάξει η δομή των μεταφορών σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό Στη δική μου τροπολογία έκανα κάποιες αλλαγές, ε, διότι είδα ότι προκαλούσε ε, ε, παρανοήσεις. Όλα τα οχήματα λοιπόν θα πρέπει να έχουν ταχογράφο. Ξέρουμε ότι η 3,5 τόνοι Ε, είναι το όριο των οχημάτων, ε, στους οποίους, ε, των οχημάτων στα οποία στοχεύει η συγκεκριμένη έκθεση. Η Επιτροπή Μεταφορών και η δική μας Επιτροπή προσπάθησαν να εξετάσουν αν, μπορούν, αν μπορεί να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια εάν πέσουμε κάτω από το κατόφλι των 3,5 τόνων. Υπήρξαν κάποιες ε, αντιπροτάσεις από διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, αλλά ίσως να άξιζε τον κόπο να τις εξετάσουμε αυτές, να δούμε δηλαδή ποια οχήματα προκαλούν ε, τροχαία ατυχήματα και για ποιο λόγο. Είναι μια πρόταση την οποία θα ήθελα να στηρίξω, διότι μπορεί να μην μπορούμε πάντα να έχουμε τις καλύτερες λύσεις. Ήταν τραγικό το δυστύχημα που έγινε στον περιφερειακό της Βιέννης. Τα ατυχήματα αυτά μπορεί να έχουν διάφορες αιτίες, την κούραση, την εξάντληση των οδηγών, αλλά μόλις το 0, 0,6% των ε, οχημάτων, ε, των ατυχημάτων μπορεί να οφείλονται σε κάποιες αιτίες, ε, να έχει τσακωθεί ο οδηγός, να παίρνει διαζύγιο, κακή ώρα της ημέρας. Αυτοί που οδηγούν στο χιόνι γνωρίζουν πόσο γρήγορα κουράζεται κανείς. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν τους λόγους τις αιτίε που προκαλούν την κούραση, την εξάντληση και δεν ξέρουμε και τι ποσοστό αυτών που εμπλέκονται σε δυστυχήματα είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ε, χρειάζεται λοιπόν προσεκτική ανάλυση των συνθήκων. Επανειλημμένα ε, έχουμε αναφερθεί στους καλύτερους ελέγχους. Ε, νομίζω όμως ότι το να ελέγχονται όλοι είναι υπερβολικό. Όσον αφορά τους, ε, τους δίθεν αυτοαπασχολούμενους, έχουμε... Ε, συζητήσει επανειλημμένα το θέμα, όχι σε τομεακό επίπεδο. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιόν να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του θέματος, διότι Μπορεί να αποτελεί αυτό αιτία του κοινωνικού ντάμπινγκ και της επιδείνωσης των ε, συνθήκων της, του δίκαιου ανταγωνισμού. Ανάπτυξη του φαινομένου αυτού θα προκαλούσε σημαντική ζημιά, ωστόσο δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά μόνο έναν τομέα. και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να πω. Ε, περίμενα εναγωνίως την ε, γνώμη της Κομισιόν για το κομμάτι των ε, τροπολογιών από την τροπολογία 104 και μετά, όπου προτείνεται να διατηρηθεί η οδηγία 561. Ε, δεν αναφέρθηκε σε αυτό όμως η Κομισιόν. 16 ε, Μαρτίου είναι η προθεσμία ε, για τις τροπολογίες. 28 Απριλίου στην 28 Μαΐου εξέταση στην Επιτροπή και θα πάει στη δεύτερη Ολομέλεια του Μαΐου. Ε, και θα ήθελα να τροποποιήσουμε λίγο την ημερήσια διάταξη, να πάμε ε, στην επόμενη έκθεση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα, όπως όλοι γνωρίζουν οι συνάδελφοι, άσχετα από το οποιαδήποτε οικονομία και οποιαδήποτε κατάσταση, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι. Όταν όμως συζητάμε τέτοια πράγματα μέσα σε το πλαίσιο μιας τέτοιας βαθιάς κρίσης όπως η σημερινή, όλα γίνονται πιο ευάλωτα και γι' αυτό και είναι πιο, πολύ σημαντικό να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτήν ε, την έκθεση. Εγώ θα ήθελα σύντομα να σας συνοψίσω ποια είναι η γνώμη μου και έπειτα θα το πούμε και στην Οικονομική Επιτροπή. Πρώτον, να μην θεωρήσουμε ότι ο χρόνος σταθεροποίησης La finanza come indistinto e irrilevante nelle sue ότι η, την οικονομία έτσι γενικά και αόριστα ε, θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τον αντίκτυπο. Δηλαδή, μια υπόθεση που θεωρητικά θα μπορούσαμε να κάνουμε για σημαντικές ε, και αδιάκριτες περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις για την έρευνα, για την καινοτομία και για την ε, εκπαίδευση και κατάρτιση, σίγουρα θα είχαν αντίκτυπο στη σταθεροποίηση, αλλά ταυτόχρονα θα είχαν και καταστροφικό αντίκτυπο στην ποιότητα και στην ποσότητα της οικονομικής ανάκαμψης που είναι απαραίτητη. Επίσης θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τον κοινωνικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην απασχόληση της κρίσης αυτής, ώστε να το καταστήσουμε όχι μόνο ως στόχο της στρατηγικής ε, του 2020, που θα πρέπει δηλαδή να επιληφθεί μέσω αυτής της στρατηγικής, αλλά και ως έναν στόχο της ίδιας της σταθεροποίησης. Να προσθέσω ότι θα χρειάζεται να Είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε για τον μηχανισμό της ανακατανομής των πόρων όσον αφορά τόσο τους φόρους όσο και τις αμοιβέ των ανθρώπων ώστε να μην επηρεάσουμε την αγοραστική δύναμη των οικογενειών γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις περιοριστικές και μάλιστα αρνητικές για τις συνιστώσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Έχουμε μια διαρθρωτική ανεργία μέσω και, και βράχη πρόθεσμα που θα θίγει περισσότερο τις γυναίκες, που θα θίξει μάλλον περισσότερο τις γυναίκες και άρα τα μέτρα σταθεροποίησης θα πρέπει να συνοδευτούν από μια ιδιαίτερη προσοχή που θα δοθεί στο στοιχείο αυτό οικονομικής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής. Έπειτα δεν νομίζω πως χρειάζεται να το θυμίσω, αλλά θα το κάνω παρόλα αυτά. Είναι προφανές ότι η σταθερότητα ενός ε, χρηματοπιστωτικού συστήματος περνά από το επίπεδο των εθνικών πολιτικών και από τις πολιτικές μετανάστευσης που θα πρέπει να ε, ε, αναθεωρηθούν ακριβώς ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η οικονομία ολόκληρης της Ευρώπης και των, χωρών, των επιμέρους χωρών. Θέλω να πω ότι χωρίς να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε στοχευμένες πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης και την ευ και μέσω της ε, πρόσβασης στις χώρες μας ε, αλλοδαπών που έρχονται εδώ να δουλέψουν αλλά δίνοντάς τους την ιδιότητα του πολίτη δύσκολα μπορούμε να σκεφτούμε όντως ανάπτυξη και το ίδιο δύσκολα θα βρούμε και την ποσότητα πλούτου ώστε να δώσουμε κοινωνική ανακούφιση από τη μία πλευρά και πρόνοια και από την άλλη να εγγυηθούμε και την οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια και κοινωνική πρόνοια που είναι η βάση για την ε, συνοχή μέσω της χρήσης των πόρων που διαθέτουν τα κράτη για τις πολιτικές αυτές. Σίγουρα θα είναι αυτό στην καρδιά της στρατηγικής 2020 για την οποία πιστεύω πως θα πρέπει να υπάρξει ένα σύμφωνο για την οικονομική, ε, ε, την κοινωνική πολιτική αλλά και την πολιτική απασχόλησης που θα ξεκινά από τα όσα έχει ήδη ορίσει η Ευρώπη για τον κοινωνικό διάλογο και την ε, ευέλικτη ασφάλεια, αλλά και θα εισάγει όπως θα πρέπει ένα σύστημα το οποίο θα βραβεύει όποιον φέρεται αποτελεσματικά και κατάλληλα και θα τιμωρεί αντίθετα εκείνον που δεν δέχεται ή που δεν σέβεται τους ε, βασικούς προσανατολισμούς. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαστεί μέγα συντονισμός, όχι μόνο κατάλληλες ρυθμίσεις. Και θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί η πολιτιστική δυνατότητα αλλά και αυτά όσα μπορούν να προσθέσει, μπορεί να προσθέσει η πράσινη οικονομία στην παραδοσιακή μεταπητική βιομηχανία που έχει χαρακτηρίσει εδώ και δεκαετίες το δικό μας ε, κόσμο. Και επίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι η χρήση των πόρων που θα δώσει σταθερότητα θα πρέπει να γίνει δίκαια και ισόρροπα. Γι' αυτό και θα είναι πολύ σημαντικό το πράσινο βιβλίο για το σύστημα το συνταξιδοτικό της κάθε χώρας. Πιστεύω πως ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός δρόμος θα είναι να διατηρηθούν τα δημόσια συστήματα που χαρακτηρίζονται από ισότητα και δικαιοσύνη, όπου όμως θα προσθεθούν στο δεύτερο πυλώνα ε, εκείνο το το ιδιωτικό κομμάτι, όπως θέλετε το λέτε, ε, ε, έτσι ώστε όσα δεν μπορούν να τα εγγυηθούν τα κράτη να, να τα εγγυώνται ενδεχομένω η συμβατική αποταμίευση, δηλαδή η, ε, τα ασφάλιστα τα οποία θα μπορεί να δίνει προσωπικά κάθε άνθρωπος ώστε να διασφαλίσει το μέλλον του δηλαδή συνδυασμό ιδιωτικού με δημόσιο τομέα, ώστε να διατηρηθούν τα στοιχεία προστασία και συνοχής που μέχρι τώρα τέλεσαν μια από τι βάσεις ε, του, του, του συστήματος πρόνοιας στις ιστορικές του συνιστώσεις και σε όλες τις εμπειρίες που χαρακτηρίζουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, νομίζω πως θα πρέπει πολύ να προσέξουμε όλα τα θετικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από την μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Βέβαια η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα είναι διαφορετική για ιστορικούς λόγους αλλά και λόγω της παγιωμένης κατάστασης σε κάθε χώρα. Αλλά είναι προφανές πως ε, μια διαφορετική διοργάνωση των ε, δραστηριοτήτων και των ε, διοικητικών δομών των ε, τοπικών και εθνικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές ε, εξοικονομήσεις ε, εισάγοντας όχι μόνο παραγωγικότητα στην εργασία και ποιότητα αλλά επίσης επιτρέποντας από τα εξοικονομήσεις σημαντικές που αν προσθεθούν στις υπόλοιπες θετικέ δράσεις θα οδηγήσουν στο να φτάσει σύντομα η οικονομία με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα επίπεδα σταθερότητας που είναι απαραίτητα. Νομίζω πως αυτές είναι βασικά οι παρατηρήσεις που θα πρέπει να απευθύνουμε προς την Οικονομική Επιτροπή που είναι επί της ουσίας αρμόδια για την έκθεση αυτή και είναι εξάλλου παρατηρήσεις οι οποίες προκύπτουν από τις συζητήσεις που κάναμε μεταξύ μας και από την ε, δουλειά που έχει κάνει η Ειδική Επιτροπή για την Οικονομική Κρίση και που αρχίζει να χαράζει κάποιες γραμμές, τουλάχιστον όσον αφορά τις προτεραιότητες. Αυτά ήθελα να σας πω και ε, όσον αφορά τις τροπολογίες, ε, θυμήσατε Πρόεδρε πως ε, έχουν μειωθεί, είναι λίγες, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει, ούτε μας εμποδίζει τη δυνατότητα να κάνουμε μεταξύ μας αποδοτική εργασία που να είναι χρήσιμη κυρίως για την Επιτροπή που θα λάβει τη γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γεζιβιέρσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου, αν μου επιτρέπετε, για την έκθεση του κυρίου Κομφεράτη. Στην πρώτη παράγραφο λέγει ο εισηγητής ότι η αύξηση της ανεργίας και η αύξηση του χρέους δεν επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη, τη μεγέθυνση της οικονομίας. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό. Η ε, ανεργία επιβαρύνει πάρα πολύ τον προϋπολογισμό κάθε χώρας. Στη δεύτερη παράγραφο λέγει ε, κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνη. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για αναζωγόνηση της οικονομίας και της βιομηχανίας, αλλά για επενδύσεις παραγωγικές που να βοηθούν την ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε, να προωθούμε την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και με επενδύσεις για να έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας. Και είναι πολύ μεγάλο εδώ το δυναμικό. Σε ό,τι αφορά το σημείο 5 της πρότασης του κ. Κομφεράτη πάντα, Εκεί αναφέρεστε ε, σε μια σωστή μεταναστευτική πολιτική. Οι εμπειρογνώμονες μας λέγουν ότι η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να καλύψει το δημογραφικό έλλειμμα που συνδέεται με τη γύρανση της κοινωνίας. Και ε, ακριβώς και η πολιτική μετανάστευση θα πρέπει εκεί να εστιάζεται. Δηλαδή τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει στην Ευρώπη. Απασχόληση δηλαδή προσώπων και άνω των 50 ετών ή και των νέων. Στην παράγραφο 7 επίσης μιλάτε για την αναδιανομή των πόρων. Και θέλετε να διατηρήσετε τουλάχιστον το σημερινό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Πρέπει να βρούμε νέους πόρους, ειδικά για τις συντάξεις, ε, γιατί ε, δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται τόσο πολύ ο δημόσιος κορβανάς. Και μιλάτε και για δύο πυλώνες ε, για την μεταρρύθμιση των συντάξεων. Εγώ θα ήθελα και ένα τρίτο πυλώνα, δηλαδή και ένα σύστημα κεφαλαιοποίησης να μπορούν να αποταμιεύουν οι εργαζόμενοι μισοτοί για τη σύνταξή τους και έτσι θα επιβαρύνεται λιγότερο το κράτος. Και έρχομαι στο σημείο 9 τώρα. Ε, αναφέρεστε στην προοδευτικότητα της φορολογίας ε, για την καταπολέμηση της φτώχειας και για περισσότερη συμπερίληψη στην κοινωνία και λιγότερο κοινωνικό αποκλεισμό. Εγώ θεωρώ ότι η φορολογική πολιτική θα πρέπει να είναι μάλλον πιο ισόρροπη με βέλτιστη χρήση των πόρων από τους φόρους για να μην έχει μεγάλο μισολογικό μη μισολογικό κόστος και η εργασία για να δημιουργούμε νέες θέσεις απασχόλησης και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας στην Ευρώπη. Ο εισηγητής επίσης δεν αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι οι εισφορές, οι κοινωνικές εισφορές. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να ακολουθούν την ίδια μέθοδο ε, στην υποβολή των ε, εκθέσεών τους. Επίσης, κάτι άλλο που δεν βλέπω είναι καμία αναφορά δεν έχετε στην πολιτική υγείας, γιατί και αυτή καταναλώνει πάρα πολύ δημόσιο χρήμα. Καλή ε, υγεία, καλύτερη όμως η πρόληψη. Γιατί θέλουμε οι πολίτες να εργάζονται και μετά την ηλικία των 65, αλλά με καλή υγεία και να τους το επιτρέπει και η υγεία τους αυτό. Για παράδειγμα, οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι οι Βρετανοί, ως παράδειγμα, σε προχωρημένη ηλικία πάσχουν από αμνησία και σε λιγότερη προχωρημένη, από τα 40 και πάνω. Επίσης, δεν γίνεται λόγος κανένας για τη δημόσια εκπαίδευση και αυτό πολύ σημαντικό, το κόστος της εκπαίδευσης. Ε, αυξάνεται ε, συνεχώς σήμερα. Δεν έχουμε καλό σύστημα εκπαίδευσης. Σήμερα στην Ευρώπη δεν ε, μορφώνουμε ε, δημιουργούς, δεν εμπνέουμε, καταρτίζουμε κάποιους ανθρώπους που καλούνται να εφαρμόσουν πράγματα που άλλοι έχουν εφεύρει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα ολίγα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να σας ενημερώσω ότι Προθεσμία της τροπολογίας είναι 6 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, ήδη έχει ανακοινωθεί. Ε, συζήτηση του σε 16 Μαρτίου, ε, υιοθέτηση στην Επιτροπή 17 Μαρτίου, υιοθέτηση στην ΕΚΟΝ 17 Απριλίου και υπολογίζεται να συζητηθεί στη δεύτερη ολομέλεια του Μαΐου στο Στρασβούργο. Ε, δεν νομίζω ότι έχει έρθει ακόμα ο Ρίτσαρτ Χάουιτ. Μήπως είναι δυνατόν λοιπόν να ε, συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Σέρκας να σας ενημερώσω όμως επίσης ότι ίσως ε, να ψηφίσουμε γύρω στις 5. Παρακαλώ ενημερώστε ε, όλα τα μέλη των πολιτικών σας ομάδων, ε, μπορεί πιο νωρίς, πιο αργά. Απλά να το γνωρίζετε παρακαλώ. Αν μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στην έκθεση του κυρίου Σέρκα, για την ενιαία διαδικασία υποβολή αίτηση για τη χωρίς του υποκόου τρίτων χωρών ενιαία άδεια διαμονή και εργασία στην επικράτεια κράτου μέλου και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για του εργαζομένου τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτο μέλο. Παρακαλώ, κύριε Σέρκα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς Σήμερα αρχίζουμε μια συζήτηση για ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ σημαντικό που θα απαιτήσει βεβαίως πολύ πιο συγκεκριμένα σχόλια από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω λίγο το γενικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει μια οδηγία σχετικά ε, με την ενιαία άδεια διαμονή και ε, τα δικαιώματα που έχουν οι μετανάστες και οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι πολύ ευρύτερο το πλαίσιο ε, για τη μετανάστευση τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία πολλά χρόνια το ζητούμε. Και το ζητούμε με όρους πάρα πολύ ξεκάθαρους. Για ποιο λόγο. Πρώτον, για να απλουστεύσουμε τα διοικητικά εκείνα στοιχεία που θα επιτρέψουν να έχουμε μια ενιαία διαδικασία για άδεια διαμονής και εργασίας, να είναι πολύ πιο εύκολο να καλύπτονται οι ανάγκες εργατικά χέρια που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε δικαιώματα στους νόμιμα διαμένοντες ε, πολίτες τρίτων χωρών για διάφορους στόχους. Καταρχάς θα πρέπει βεβαίως να τους μεταχειριζόμαστε ως πρόσωπα, ως ανθρώπους αλίμονο που έχουν ε, αντίστοιχα δικαιώματα με εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι περισσότερο τώρα, αυτή τη στιγμή. Γιατί από το έτος 2004, που ήταν το πρώτο πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους ε, νόμιμους και παράνομους εργαζομένους μετανάστες και ε, είναι ευρία η συνένεση ότι θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι κατά της λαθρομετανάστευσης και πάρα πολύ γενναιόδοροι από την άλλη για την ένταξη στην κοινωνία και την ενσωμάτωση της νόμιμης μετανάστευσης. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μια πολιτική που να διέπεται και από τα δύο αυτά. Έτσι. Να είμαστε πραγματικά αμήλικτοι ανελέητη με τη λαθρομετανάστευση, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε εκείνοι που μπαίνουν νόμιμα στην Ευρώπη να έχουν ένα πλαίσιο και μια νομική ασφάλεια και δικαιώματα για να μπορούν να εντάσσονται πραγματικά στις κοινωνίες μας. Επιπλέον, και θέλω να τονίσω, αυτές οι δύο πολιτικές ε, αλληλεπιδρούν. Όταν γίνεται λόγος για το μαγνήτη, την προσέγγιση της λαθρομετανάστευσης, έρχονται πάρα πολλοί ε, υπήκοοι τρίτων κρατών ακριβώς με συνθήκες που δεν σέβονται τον νόμο. Όταν έχουμε μια μαύρη ε, εργασία χωρίς δικαιώματα, με πλήρη έλλειψη ε, νομικές ασφάλειας και κάλυψης, αυτό τραβάει τη λαθρομετανάστευση και αυτό πολλαπλασιάζει τους δουλέμπορους και τις μαφίες. Αντίθετα, αν έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μονίμων και νομίμων μεταναστών, τότε καταπολεμούμε ταυτόχρονα και τη λαθρομετανάστευση. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα πάει στην Ευρώπη και θα βρει δουλειά στη μαύρη και χωρίς δικαιώματα και χωρίς υποχρεώσεις. Θα ξέρουν ότι θα καλύπτονται πάντα από κοινωνική νομοθεσία οι εργαζόμενοι και οι μετανάστες. Σιγά σιγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν διαφαίνεται μια νοοτροπία, μια κουλτούρα που προσπαθεί ταυτόχρονα να, απαντήσει και στο δικαίωμα των ανθρώπων αυτών αλλά και σε μια ανάγκη της υπήρου μας. Χρειαζόμαστε ε, κανόνες και δικαιώματα για τους ανθρώπους αυτούς που επαναλαμβάνω διαμένουν νόμιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2007 έχει εξαγγείλει την οδηγία αυτή ως οδηγία πλαίσιο που θα ε, ρύθμιζε την ενιαία διαδιαμονής και εργασίας αλλά και το σύνολο των δικαιωμάτων που θα έχουν όλες οι κατηγορίες εργαζομένων. Βέβαια από εκεί και πέρα επιμέρους ε, εξήγηλαν και ξεχωριστές οδηγίες για κάθε κλάδο εργαζομένων. Σήμερα σε αυτή την πρόταση οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, ανακαλύπτουμε ότι η συζήτηση δεν θα είναι ούτε εύκολη μεταξύ μας, αλλά δεν θα είναι και εύκολη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Πρώτον, δεν θα είναι εύκολη συζήτηση. Γιατί? Η αιτιολογική έκθεση λέει ότι θα είναι η οδηγία πλαίσιο που θα συγκεντρώνει εγκάρσια οριζόντια τα δικαιώματα όλων των ξένων εργαζομένων, εκτός από εκείνους που έχουν ε, άδεια μακράς διάρκειας. Αυτή η οδηγία θα έπρεπε να ε, έχει φτάσει νωρίτερα από τις επιμέρους, τις τομεακές και τις κλαδικές, αφού είπαμε ότι είναι οδηγία πλαίσιο. Εάν θέλουμε να έχουμε απουσία αντιφάσεων και συνοχή που θέλουμε και το απαιτούμε, θα έπρεπε αυτή η οδηγία που λέει ότι είναι πλαίσιο να έρθει πριν από κάποιες άλλες για κυρώσεις, ας πούμε, ε, προς επιχειρηματίες ή ε, για την ε, εξειδικευμένη εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε έτσι ώστε η οδηγία αυτή να ξαναγίνει εγκάρσια, παρόλο που ήρθαν προηγουμένως οι κλαδικές ή τομεακές οδηγίες και δεν είναι καθόλου λογικό αυτό. Παρά τα αντίθετα που είχε δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν ήδη επιμέρους κείμενα ε, τα οποία έχουν ε, λάβει την ε, νομοθετική οδό. Και υπάρχουν και άλλες οδηγίες στο κοινοτικό και εκτιμένο όπως είναι ε, η οδηγία ε, για το νομοθετικό πλαίσιο για τους εργαζομένους μακράς διάρκειας, εκείνους που είναι στην Ευρώπη εδώ ε, ως ε, υπότροφοι, ως σπουδαστές ή με ανταλλαγή εδώ ή κάνουν έρευνα επιστημονική είτε θελοντική άμυστη εργασία. Όλα αυτά λοιπόν είναι δύσκολα. Και η πρώτη αυτή δυσκολία είναι εκείνη που σας είπα. Ότι θέλουμε να είναι οδηγία πλαίσιο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρξει συνοχή. Γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίει τις γενικές αρχές με τις επιμέρους απαντήσεις. Αυτή ήταν η πρώτη δυσκολία. Έχουμε και μια δεύτερη που θα πρέπει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Είναι ότι η οδηγία αυτή έρχεται στο Κοινοβούλιο με τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας της δικής μας Επιτροπής με την Επιτροπή Ελευθεριών. Εγώ δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ ποιος έχει εφεύρει εδώ τους κανόνες στο Κοινοβούλιο, αλλά ο κανόνας και οι κανονισμοί του Κοινοβουλίου κινδυνεύουν να μας κάνουν να χάσουμε την ε, ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Μιλάμε για τέσσερις αιτιολογικές σκέψεις και για τρία άρθρα. Πώς θα το κάνουμε αυτά. Ε, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελευθεριών. Εμάς μας πέφτει μια παράγραφος ενός άρθρου και εκείνοι θα εξετάσουν όλα τα άρθρα. Η οδηγία αυτή έχει δύο ξεχωριστά κομμάτια, το ένα αναφέρεται στη διαδικασία και το άλλο στα δικαιώματα. Και διασταυρώνονται και στις δύο περιπτώσεις οι αρμοδιότητες των δύο επιτροπών. Ούτε καν έχουμε επιμέρους ε, αρμοδιότητες με τρόπο σαφή. Διασταυρώνονται ακόμα και οι αρμοδιότητές μας. Έτσι λοιπόν, όπως ήταν λογικό, εγώ θα ζητήσω τροπολογίες για τις αιτιολογικές σκέψεις και το τμήμα των άρθρων που είναι δική μας αρμοδιότητα. Αλλά και ο εισηγητής σας και οι βουλευτές ε, έχουν δυσκολία να μην κάνουν τροπολογίες και σε άλλα άρθρα έστω και γνωμοδοτικά, για αυτά που κάνει η Επιτροπή Ελευθεριών. Γιατί αναπόφευκτα, πώς να το πω, θα χρειαστεί να υπάρξει μεγαλύτερη ε, συνοχή. Γιατί ήρθε ένα διοικητικό μαχαίρι και έκοψε στα δύο τη δουλειά ανάμεσα στις δύο επιτροπές, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρος αυτός ο διαχωρισμός. Επί της ουσίας τώρα, θα πρέπει να κάνουμε μια ε, εκβαθέων πολιτική συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο κοινοβούλιο εμείς τι κάνουμε εδώ. Ερχόμαστε να συμπληρώσουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέει στην αιτιολογική έκθεση το κείμενο της Επιτροπής ότι είναι μια οδηγία που εκτός από τα διοικητικά θέματα θα δημιουργήσει και μια νομική ομπρέλα για να εγγυάται δικαιώματα, ελευθερίες, δίκαια μεταχείριση και ισότητα στη μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων που έρχονται από τρίτες χώρες και των δικών μας, ε, των πολιτών της Ένωσης. Αυτά, αγαπητή Πρόεδρε, τα λέει όμως στην αιτιολογική έκθεση. Στο διατακτικό έρχεται να γκρεμίσει όλα αυτά που λέει η αιτιολογική έκθεση. Ε, πρώτον, με ένα άρθρο 3, όπου γίνεται λόγος για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αφήνει απ' έξω ομάδες που θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ. Σπάει δηλαδή τη λογική της οδηγίας. Για παράδειγμα, αν βγουν εκτός οι εργαζόμενοι εποχιακοί στην Ευρώπη. Μα μιλάμε για ίσα δικαιώματα, για ίδια δικαιώματα για αυτούς που εργάζονται εδώ. Αλλά οι εποχικοί τι γίνονται είναι από εκείνους που εργαζόνται ε, και χρειάζονται πολύ περισσότερη προστασία. Για να σπάσει η λαθρομετανάστευση. Γιατί ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη θα πρέπει να υπόκειται στην εργατική νομοθεσία και στην κοινωνική νομοθεσία και την κοινωνική ασφάλιση στα κράτη-μέλη. Ε, πώς μπορούμε να πούμε με τέτοιο τρομερό τρόπο αυτή την αντίφαση μεταξύ των όσων λέει η αιτιολογική έκθεση και τα άρθρα. Ενδεχομένως, ενδεχομένως και μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο, κάποια διέξοδο να πούμε ότι υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία. Δεν υπάρχει όμως ακόμα. Δεν έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο πρόταση οδηγίας για τους εποχικούς εργαζομένους. Και αν μη τι άλλο και ήδη σας λέω από τώρα τι θα συζητήσουμε, μέχρι να έρθει δική νομοθεσία, αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπουν στην οδηγία αυτή, να καλύπτονται. Και δεν ξέρω επικουρικά, συμπληρωματικά, παραπληρωματικά από την οριζόντια αυτή νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και με τους εργαζομένους που αποσπά ε, μια επιχείρηση προς την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς είναι δυνατόν να μην καλύπτονται υποχρεωτικά. Και πόσο κατάφορη είναι αυτή η αντίφαση ανάμεσα στο κείμενο και τις προθέσεις και τις εξαγγελίες για την οδηγία αυτή. Τελευταίο, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλέσω τους συναδελφούς να μελετήσουν σε βάθος, ε, γιατί το θέμα αυτό υπάρχει και άλλη τεράστια δυσκολία στο άρθρο 12 που είναι πλήρης δικήμα δικαιοδοσία, στο πρώτο άρθρο αναφέρονται δικαιώματα για την κοινωνική ασφάλιση, για την απασχόληση, για την παιδεία, για τα δικαιώματα τα κοινωνικά και τα εργασιακά και στο δεύτερο ε, τμήμα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να αποκλίνουν, να εξαιρεθούν από ορισμένα δικαιώματα. Μα είναι πάρα πολύ αμφίβολο αν μπορεί κάποιος που ε, εργάζεται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην απολαμβάνει αυτών των δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν, για το πεδίο εφαρμογής ε, προκύπτουν διάφορα γιατί αφήνει χωρίς νομική κάλυψη πολλές κατηγορίες εργαζομένων αλλά ακόμα και αυτοί που καλύπτονται από το άρθρο 3 στο 12 μπορεί να ε, εξαιρεθούν επειδή έτσι θα επιθυμεί κάποια χώρα μέλος. Θα πρέπει να δούμε την ε, πραγματικότητα. Πρόκειται για οδηγία. οδηγία. Σέβεται τα διαδικαστικά και μάλλον ως προς τα διαδικαστικά είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά για το αν θα δημιουργήσει ένα αρμονικό νομικό σύλλογο είναι πάρα πολύ αφισβητήσιμο αυτό και συζητήσιμο και ελέγχεται. Ε, συμπέρασμα, συνάδελφοι, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Τα θέματα αυτά δεν είναι καθόλου απλά. Είναι πάρα πολύ επίκαιρα, πάρα πολύ επίκαιρα. Όχι μόνο για να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για την νομική, νόμιμη μετανάστευση στην Ευρώπη, αλλά για να γίνει πραγματικότητα αυτό που χρόνια ολόκληρα πρεσβεύουμε και υποσχόμαστε και στους δικούς μας πολίτες και στους πολίτες τρίτων κρατών, ότι θα είμαστε αμήλικτοι και πάρα πολύ απαιτητικοί απέναντι στη λαθρομετανάστευση, αλλά αυτοί που διαμένουν νόμιμα στην Ευρώπη θα έχουν ε, αντιμετώπιση ως άνθρωποι ε, με δίκαιο τρόπο και με ίση μεταχείριση με τους δικούς μας πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes, thank you. Uh, thank you very much for that. Uh, yes, I know how difficult it is when you're... Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι όταν προσπαθεί κανείς να μοιράσει ευθύνες, πιανού ευθύνη το κάθε άρθρο, ξέρω, το ίδιο είναι και με την οδηγία κατά των διακρίσεων, αλλά η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών το συζητά σήμερα και γι' αυτό και δεν έχουμε κανέναν από την Επιτροπή να το συζητήσει μαζί μας αυτή τη στιγμή. Αλλά προφανώς θα συναντηθείτε και με την Επιτροπή Πολιτικών ε, ε, Ελευθεριών εφόσον είναι υπό τη διαδικασία Hughes για να δούμε αν μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες σε αυτή την έκθεση. Γιατί εγώ αυτό έκανα με την οδηγία κατά το διακρίσεων. Αλλά θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι αν προσπαθήσουν να τροποποιήσουν οποιασδήποτε παραγράφους που δεν είναι δική μας ευθύνη, τότε αυτό θα θεωρηθεί ε, ως μη αποδεκτό. Να σας δώσω και το χρονοδιάγραμμα, λοιπόν για την προθεσμία είναι 24 Απριλίου το μεσημέρι, ε, Μαρτίου συγγνώμη, το μεσημέρι, υιοθέτηση της έκθεσης ε, στις 28 Απριλίου και ταυτόχρονα και στην Επιτροπή επί της και Μάιος για την Ολομέλεια. Αν τροποποιήσετε λοιπόν τροπολογίες που δεν είναι δική μας ευθύνη, θα θεωρηθούν μη αποδεκτές από τη γραμματεία του Κοινοβουλίου. Ο κύριο Χάουιτ έχει καταφτάσει. Οπότε να επανέλθουμε σε εκείνο το σημείο τη τη διάταξη που αφορά σε κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ και τα ανθρώπινα δικαιώματα στι διεθνεί στις διεθνείς συμφωνίες. Κύριε Χάουιτ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας συγχαίρω. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρατε να φτάσετε από τη West Midlands, δεν ξέρω αν χιόνιζε ή όχι. Μπράβο σας πάντως που είστε εδώ. Και ευχαριστώ που ήσασταν και ευέλικτοι με τη μυρίσια διάταξη σήμερα. Μου ζητήθηκε λοιπόν να κάνω μια γνωμοδότηση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Είναι πολύ ευρύ ε, ε, τομέας. Ήδη συντάσσουμε γνωμοδότηση. Η βασική έκθεση είναι στην Επιτροπή Εμπορίου και έχει γίνει δημόσια συζήτηση εδώ και χρόνια για το πόσο συνδέουμε τις προδιαγραφές του κοινωνικού ε, και του περιβαλλοντικού τομέα με τον ΠΟΕ, το Παγκόσμιο Οργανισμό για το εμπόριο, ο καθένας έχει την άποψή του εδώ και είναι δύσκολο να μπορέσουμε να κατασταλάξουμε ε, σε λίγες παραγράφους ε, και έκανα ό,τι μπορούσα. Καταρχήν λοιπόν στην πρώτη παράγραφο για να σας πω πρακτικά πώς έχει το, η δική μου γνωμοδότηση παρουσιάζω ποια πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι οι αρχές μας. Δηλαδή απορρίπτουμε τον προστατευτισμό ή οποιαδήποτε απόπειρα να, να παρέμβουμε στις ε, νόμιμες ε, διεκδικήσεις κάθε χώρα και την ε, κυριαρχία της αλλά ότι μπορούμε να επηρεάσουμε μέσω των εμπορικών συμφωνιών και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να υποστηριχθεί από το όλο το πολιτικό φάσμα της Επιτροπής και έπειτα αντί να προσπαθήσω με έτσι πιο γενικό τρόπο να αντιμετωπίσω το θέμα, με διάφορες σαρωτικές δηλώσεις. Έχω προσπαθήσει να φτιάξω μια γνωμοδότηση πολύ πρακτική και ρεαλιστική, λεπτομερής όσον αφορά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες. Και βέβαια εδώ είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης και γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε τη γνωμοδότησή μας στις κοινωνικές προδιαγραφές και τις σχέσεις με το Διεθνή Οργανισμό για ε, την ε, Εργασία. Έχω διάφορε συστάσει λοιπόν. Παράγραφο 1 αφορά την ερμηνεία που χρησιμοποιεί ο ΠΟΕ στο άρθρο 24 όπου λέει ότι υπήρξε ιδιαίτερα ζηλότυπη ερμηνεία αυτή του άρθρου και ότι θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την προστασία ευαίσθητων τομέων είτε εντός Ευρώπης είτε εκτός. Στη δεύτερη παράγραφο Βλέπουμε τι συμβάσει πυρήνα του διεθνού Γραφείου εργασία, τις γνωρίζουμε αυτές, αλλά από το 1998 υπήρξε μια σειρά οκτώ βασικών συμφωνιών, συμβάσεων μάλλον, που το διεθνέ Γραφείο εργασία θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ άσχετα από το τι έχει επικυρώσει η μεμονωμένη χώρα, συμπεριλαμβανομένη ε, τη ελευθερία του συνεταιρίζεστε, για παράδειγμα. Αυτό που λέμε είναι ότι η πραγματική επικύρωση και εφαρμογή αυτών των ε, βασικών ε, συμβάσεων θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και των εμπορικών της συμφωνιών και θα πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο επίπεδο και με το ίδιο καθεστώς όπως και οι πρόσβαση στην αγορά. Πράγμα το οποίο πολύ ισχυρίζονται δεν ισχύει τώρα. Στην τρίτη παράγραφο λέω ότι η Κομισιόν βασίζεται υπερβολικά πολύ στα διεθνή σώματα και στι διεθνεί συνθήκε. Δεν ξέρω αν εδώ και ε, ανακούνε, κανονικά είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εδώ. Εδώ δεν θέλω να επικρίνω την Επιτροπή. Απλώ πιστεύω ότι τώρα λόγω τη αυξανόμενη περιπλοκότητα του παγκόσμιου εμπορίου ε, Επίση, με τη στροφή της Ευρώπης για να έχει περισσότερες διμερεί συμφωνίε σε μια φάση όπου έχει ήδη παρέλθει η εποχή όπου βασιζόμασταν στους διορυθμίους οργανισμούς για να το κάνουν αυτό ε, ε, εξ ονόματός μας. Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε τη δυνατότητα στην Ευρώπη να προβαίνουμε στις δικές μας κρίσεις για το σε ποιο βαθμό οι διάφορες χώρες ε, τήρουν τις προδιαγραφές για την βιώσιμη ανάπτυξη. Έπειτα στην παράγραφο 4 ζητώ να εξετάσουμε τον κανονισμό GSP, δηλαδή τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά που δίνουμε σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών για την Ευρώπη, γιατί υποτίθεται ότι συμμορφούνται προς τις συμβάσεις αυτές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και εδώ πολλοί είπαν ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται όλα αυτά είναι, δεν είναι καθόλου συνεπή ούτε αντικειμενικά όπως θα έπρεπε. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, υπάρχουν ωστόσο και καταγγελίες και παράπονα ότι δηλαδή τα κριτήρια αυτά είναι κάπως αυθαίρετα και ότι ε, καθώς θα αναθεωρηθεί ο σχετικός κανονισμός, αυτές οι αδυναμίες θα πρέπει να ε, ξεπεραστούν, πράγμα που θα συμβεί σύντομα. Επίσης γνωρίζω πως ε, έγινε, λήφθη μια πρόταση για να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία ευνοϊκής πρόσβασης με την Σρι Λάγκα είναι ένα θετικό παράδειγμα όπου η Ευρώπη όντως ενήργησε, έδρασε. Κανείς δεν θέλει να το κάνει αυτό έτσι με ποινικό τρόπο. Θέλουμε να λειτουργήσει ως κίνητρο ώστε η χώρα αυτή να ε, τηρήσει και να, να συμμορφωθεί προς υψηλότερες προδιαγραφές. Θα δείχνει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να γίνεται με συνέπειες ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, οι, αξιο... οι... μελέτες αξιολόγησης είναι ένα καλό όχημα, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως θα έπρεπε, ώστε να επιστήσουν την προσοχή μας στο γεγονός πως όντως έχουμε ίδια ε, οικονομικά και κοινωνικά αιτήματα και ανάγκες από ευρωπαϊκή άποψη. Δεν πρόκειται για προστατευτισμό, αλλά για τα θέματα τομείς όπου υπάρχει μια πολύ γρήγορη παρακμή, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο ύφεσης, ότι υπάρχει δηλαδή μια, υπάρχουν αρχές στην εμπορική μας πολιτική και τις αναγνωρίζουμε και δίνουμε την κατάλληλη ανταπόκριση. Αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι αν λαμβάνουμε αποφάσεις από μια πλευρά μέσα στις εμπορικές συμφωνίες θα έχουν ε, αρνητικά και σε επιπτώσεις στην αναδιάρθρωση και θα πρέπει αυτά να συντονιστούν με τον ε, ε, Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί όσο θα μπορούσε. Παράγραφος 7 αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάγκη της ίδιας ε, της ε, των, διαφόρων μάλλον βιομηχανικών κλάδων να σεβαστούν τις οικονομικές και κοινωνικές προδιαγραφές καθώς και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. α πούμε, ο ΣΑ, Διεθνές Γραφείο Εργασίας και ο ΙΕ εργάζονται για τη θέσπιση ενός κοινού σετ, ενός κοινού συνόλου προδιαγραφών και ότι όλα αυτά θα πρέπει και εμείς να τα παροτρύνουμε από πλευρά των δικών μας ευρωπαϊκών πολιτικών για το εμπόριο. Και στη συνέχεια στην παράγραφο 9, γιατί στην 8 δεν θα αναφερθώ. Αναφερόμαστε σε θέματα της προσωρινής κίνησης, μετακίνησης των εργατικών χεριών σε συμφωνία με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ξέρουμε ότι αυτό έχει υπάρξει πρόβλημα εδώ στην Ευρώπη ήδη ε, με τα δικά μας δικαστήρια ανάμεσα στις δικές μας χώρες και αν δεν το προσέξουμε θα υπάρξει πρόβλημα μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών και γι' αυτό και ζητώ να αποφευθεί και να καταστεί σαφές πως σεβόμαστε τις διεθνείς προδιαγραφές εργασίας και τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις στις χώρες εταίρους. Τέλος, ζητάμε ακόμη από τον ΠΟΕ να εξετάσει το θέμα της ερμηνείας, γιατί θεωρούμε πως ο ΠΟΕ ε, είναι ο, η βίβλος και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Όχι, είμαστε μέλη του ΠΟΕ, μπορούμε να δουλέψουμε για να αναθεώρηση και σύμφωνα με τους, κανόνες, τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ υπάρχουν πολλά θέματα ερμηνείας, τα οποία είναι αμφισβητούμενα. Και η λέξη ε, ενίσχυση, ε, βοήθεια, έχει χρησιμοποιηθεί ως θηλιά ε, πολλές φορές και επιτρέπεται παραγωγή σε πολλές χώρες που δεν σέβεται οποιαδήποτε κριτήρια απασχόλησης ή κοινωνικά κριτήρια και αυτά και πάλι θα πρέπει να εξεταστούν σε επίπεδο ΠΟΕ. Ελπίζω λοιπόν πως ε, θα σας βρει σύμφωνο η γνωμοδότησή μου. Φυσικά ε, θέλω να ακούσω τι έχετε να πείτε και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας για τροπολογίες πριν φτάσουμε στη τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής ε, θέλουν να παρέμβουν, διότι υπάρχει κοινή αρμοδιότητα από τη Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο. Κύριε Μοράλες, πρώτα σας δίνω το λόγο και κατόπιν στην Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, από την ε, Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση έρχομαι. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου να διασφαλίσει την συνοχή της εμπορικής πολιτικής με όλες τις πολιτικές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπορική πολιτική και οι εμπορικές συμφωνίες είναι μέσα τα οποία θα πρέπει να συμβάλλουν σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η παράγραφοι 1 και 6 του σχεδίου γνωμοδότησης ε, αναφέρεται στα θέματα αυτά. Θέλουμε να τονίσουμε τον ε, ρόλο της εμπορικής πολιτικής για ε, τη δημιουργία ευκαιριών για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τονίζοντας ταυτόχρονα την την ανάγκη για κάποιες αλλαγές εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Κομισιόν ε, διαπραγματεύεται ε, σχετικές ρήτρε, κυρίως στα πλαίσια του κεφαλαίου για το εμπόριο και την αναπτυξιακή βοήθεια στις εμπορικές αυτές συμφωνίες. Και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, τις πολιτικές δεσμεύσεις και ε, τη δέσμευσης με τους εμπορικούς μας ε, ε, με τους εμπορικούς μας εταίρους. αυτή είναι η, η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε και δέσμευση του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006 που έχει τονιστεί έκτοτε και που έχει στηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκτενές ψήφισμα του 2007 αναφέρεται ένα πρόγραμμα εργασίας όπου αναφέρονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ο κοινωνικός διάλογος ε, και η ποιοτική στόχη. Γι' αυτό περιλαμβάνει τα λεγόμενα βασικά πρότυπα των εργαζομένων αλλά ε, το πρόγραμμα αυτό ε, περιλαμβάνει κάτι παραπάνω. Ε, θέλει να διασφαλίσει όχι μόνο κάποια ελάχιστα δικαιώματα, αλλά στοχεύει στην, στον καλύτερο συνδυασμό της οικονομικής ανταγωνιστικότητας με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και είναι σημαντικό το ελεύθερο εμπόριο να συνδυάζεται με την αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε να κερδίζουν από αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εμπορική της εταίροι. Γι' αυτό τα κεφάλαια για την αναπτυξιακή βοήθεια καλύπτουν κυρίω τρία στοιχεία. Καταρχήν, ε, καλούν η αποτελεσματική εφαρμογή των τεσσάρων ε, προτύπων ε, που αναφέρονται στι θεμελιώδει συμβάσει του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Δεύτερον, τονίζονται οι πολιτικοί στόχοι. Και τρίτον, στοχεύεται στη δημιουργία μια πλατφόρμα διαλόγου και ε, αυτές οι διατάξεις ε, στηρίζονται από συγκεκριμένα μέτρα, την ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρεται σε κυρώσεις, αναφέρεται σε θετική δέσμευση των εμπορικών μας εταίρων ε, στα κοινωνικά πρότυπα και τους κοινωνικούς στόχους, διότι η ανάπτυξη μπορεί να βασιστεί μόνο σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και στην ε, ανάπτυξη της αίσθησης της ιδιοκτησίας. Τα κεφάλαια για την αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να υπόσχονται αποτελέσματα στον στο, όσον αφορά αυτό και είναι σημαντικό η κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Να, ε, ε, ε, να έχουν αποτέλεσμα οι ρήτρε αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να σας δώσει γραπτός παρατηρήσεις για την για το σχέδιο χρονομοδότησης ε, που έχετε μπροστά σα. και ο συνάδελφό μου από την Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο θα προσθέσει κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο. Λόγω του περιορισμού του χρόνου είμαστε διατεθειμένοι να σας υποβάλουμε γραπτό στις παρατηρήσεις μας όπως και να έχει, θα θέλαμε να, με κάποια ε, παραδείγματα να σας ε, αναφέρουμε τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν πιο αναλυτικά. Θα πρέπει να ε, θυμόμαστε ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρε σε εμπορικές συμφωνίες είναι ένα πολύπλοκο θέμα και θα πρέπει να συζητηθούν προσεκτικά τα θέματα που θίγονται στη γνωμοδότηση. Ένα θέμα που θέλουμε να τονίσουμε είναι, για παράδειγμα, η ανάγκη για διάκριση ανάμεσα στους προαιρετικούς κανόνες, τα έγγραφα, κατεύθυνση κατεύθυνσης και τις δεσμευτικές ρήτρες. Ε, θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε, να διασφαλίσουμε το το δικαίωμα ε, του, του Κοινοβουλίου και άλλων να λαμβάνουν τις δικές τους ε, αποφάσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, θα ήταν, ότι δεν θα ήταν σκόπιμο κάποια κάποιες, κάποιους προαιρετικούς ε, κώδικες, ε, να τους κάνουμε υποχρεωτικούς κανόνες, όπως ε, προτείνεται στην παράγραφο 7. Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν σχεδιαστεί ως νομικά μέσα τα οποία μπορούν να επιβληθούν. Επιτέλους, επίσης, η Κομισιόν συμφωνεί ότι τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να προωθούν τις βέλτιστες εμπορικές πρακτικές, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνική ευθύνη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την τήρηση των προαιρετικών ε, κωδίκων δεοντολογίας και των ε, διεθνών ε, μέσων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μελέτες, ε, οι αξιολογήσεις ε, των επιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 ε, εκπονούνται από ανεξάρτητους φορείς, αλλά η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταλήξουν σε δική τους αξιολόγηση των πτυχών της αηφορίας στα πλαίσια κάθε εμπορική συμφωνίας. Το εάν ή όχι αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τα αποτελέσματα των ε, εμπειρογνωμόνων. Επίσης, ε, όσον αφορά την παράγραφο 4, η Επιτροπή πιστεύει ότι οι ε, εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να βασίζονται σε κάποια αντικειμενικά κριτήρια και γι' αυτό εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από τις ε, γνωμοδοτήσεις και το σύστημα ε, παρακολούθησης ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτό ισχύει και αμφισβητούμε αν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετα στοιχεία. Είναι πολύπλοκη η κατάσταση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν την τελευταία λέξη, δεν θα πρέπει να υπάρχει να γίνεται αυτόματα η εφαρμογή μηχανισμών. Χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το σχέδιο γνωμοδότησης ε, συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό ε, νομικών και τεχνικών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν αναλυτικά. Γίνεται αναφορά σε νομικές ρήτρες, ε, το άρθρο 24 του, ε, της Συμφωνίας ε, Προτιμήσεων και επίσης στα συστήματα επιδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί αναφέρονται και κάποιες συγκεκριμένες χώρες, κάποια συγκεκριμένα θέματα. Αυτά θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά από εμπειρογνώμονες, ε, θα πρέπει να συζητηθούν και εάν η Επιτροπή σας θέλει ε, σήμερα περαιτέρω ε, σχολιασμό των σημείων αυτών, είμαστε, είμαστε στη διάθεσή σας. Αλλιώς θα σας στείλουμε γραπτός τις παρατηρήσεις μας για να τις εξετάσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να πω απλά ότι ε, ε, η ψηφοφορία θα γίνει στις 5. Ε, Μία αντίρρηση ακούσαμε, αλλά δεν βλέπω κανένα λόγο να καθυστερήσουμε τις ψηφοφορίες. Οι περισσότεροι συντονιστές θέλουν να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν αμέσως μετά τη συζήτηση αυτή θα ψηφίσουμε. Κύριε Χάουιτ θέλετε να πάρετε το λόγο. Δεν ζήτησε κανείς άλλος το λόγο. Α, ένας. Δεν βλέπω, χρειάζομαι τα γυαλιά μου. Μπορείτε παρακαλώ να πείτε το όνομά σας, διότι δεν βλέπουμε την καρτέλα σας. Τζον Higgins από την ε, ομάδα Γκουε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τις προτάσεις του κυρίου Χάουιτ, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα θα πρέπει να είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να επιμένουμε ε, στις ε, εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Ε, δυστυχώς, τα στοιχεία που έχουμε από οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών από, διάφορες, και από διάφορους φορείς μας λένε ότι σε, πολλά, σε πολλές χώρες με τις οποίες έχει εμπορικές σχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα παραβλέπονται, αγνοούνται σε πολλές περιπτώσεις. Στην ε, παράγραφο 3 των προτάσεων του κυρίου Χάουιτ, αναφέρονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τις ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, πριν την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, αλλά δυστυχώς τα στοιχεία είναι ότι η γνώμη τους των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν λαμβάνεται υπόψη επαρκώς από την Επιτροπή και επανειλημμένα υποβάλλονται στοιχεία από φορείς που εκπροσωπούν ε, εργαζομένους και μικρούς παραγωγούς και ε, κατοίκους μικρών χωρών. Ε, στοιχεία υποβάλλονται λοιπόν από αυτούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν παίζουν ρόλο οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες στην Λατινική Αμερική για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι Ακόμα και πολυεθνικές κατηγορούνται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα ξέρουμε από οργανώσεις, για παράδειγμα, που αγωνίζονται για την προστασία του, του περιβάλλοντος. Στην παράγραφο 5 αναφέρεται η περίπτωση της Κολομβίας. και το γεγονός ότι ετοιμάζεται σχετική συμφωνία. Εγώ θα ήθελα εδώ να το τονίσω πολύ περισσότερο, να πούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει εμπορική συμφωνία με την Κολομβία τη στιγμή που τα πράγματα έχουν όσο έχουν, όπου η ε, δολοφονία ε, συνδικαλιστών έχει γίνει ρουτίνα. Επικρατεί ατιμορρησία και εκφοβισμός των ε, εργαζομένων που ε, αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ε, και τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Στο σημείο 6, ο κύριος Χάουετ πολύ συχνά αναφέρεται στο γεγονός ότι οι εμπορικέ συμφωνίε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση στο πλαίσιο τη οικονομική κρίση και θέλει να αποτρέψει την ε, ε, ε, ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς και των επένδων απασχόληση σε οποιοδήποτε τομέα τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Αλλά, κυρία Πρόεδρε, οι επιχειρήσεις εξαρτιόνται από την πρόσβαση σε φθηνό εργατικό δυναμικό και έχουμε την πολύ δυσάρεστη κατάσταση όπου εργαζόμενοι από διάφορες χώρες ε, στρέφονται ε, ο ένας κατά του άλλου. Έχουμε ένα δυσάρεστο παράδειγμα. Η Dell ε, απέλησε 1.700 εργαζομένους στην Ιρλανδία και η Πολωνία στήριζε τις την, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριζε την Πολωνία για, με, την κατάσταση της παραγωγής εκεί. Και κυρία Πρόεδρε, η τελευταία μου παρατήρηση είναι εξή. Ο κύριος Χάουιτ επιμένει ότι κάθε συμπερίληψη σε ε, εμπορική συμφωνία τη ε, προσωρινή κινητικότητα των εργαζομένων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με εθνικά πρότυπα ε, και τι συλλογικέ συμφωνίε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Πρέπει όμως να θέσω ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη μία απόφαση μετά την άλλη, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, έχουμε την Βάξχον Λεβάλ, Έχουμε την, μια απόφαση της ε, Βόρειας ε, Σαξονίας, του Λουξεμβούργου. Ε, οι αποφάσεις αυτές κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Και επιτρέπει στους υπεργολάβους να απασχολούν ανθρώπους από τρίτες ε, χώρες ε, σε πολύ χαμηλούς μισθούς και με πολύ ε, κακές συνθήκες. Θα παρακαλούσα τον κύριο Χάουιτ να σχολιάσει το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά τη λεγόμενη ερμηνεία των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε, οι αποφάσεις του δικαστηρίου σημαίνουν ότι το σημείο 9 του κυρίου Χάβερτ δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αντιδράσω σε σχέση με αυτό που, είπε, ε, που υπόθηκε για την Κολομβία. Την περασμένη εβδομάδα ως μέλος της αντιπροσωπείας ε, των σοσιαλιστών στην Κολομβία στην ε, διερευνητική των πραγμάτων επιτροπή. Και αυτό που είπε ο σα δεν ισχύει. Δυστυχώς, όλη η πληροφόρηση που έχουμε από την Κολομβία και όλες οι γνωμοδοτήσεις που ε, παίρνουμε για τα γεγονότα στην Κολομβία ε, είναι μονόπλευρε και μονομερείς. Εμείς πήγαμε στην Κολομβία, είδαμε τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό εισαγγελέα, εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολλούς συνδικαλιστές. Και εγώ ο ίδιος συνδικαλιστής είμαι και ποτέ δεν θα αμφισβητούσα αυτό που μας ε, λένε τα συνδικάτα αν δεν ήταν ε, γεγονός. Η εικόνα που μας δίνουν ε, για την Κολομβία είναι στρεβλή. Δεν ισχύει αυτό. Έχουν γίνει δημοκρατικά βήματα στη χώρα. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Τώρα εφαρμόζεται και ένας καινούριος νόμος όπου θα θεωρείται γενοκτονία η δολοφονία συνδικαλιστών. Δεν είναι εθνικό άθλημα το να δολοφονούν συνδικαλιστές στη Γολομβία όπως συχνά ισχυρίζονται κάποιοι. Ε, το γεγονό ότι τους δολοφονούν δεν έχουν να κάνουν με το ότι είναι συνδικαλιστές παρακολουθούνται ε, και ε, προστατεύονται 1.500 συνδικαλιστές. Και θα παρακαλούσα πριν κάνουμε γνωμοδότηση, πριν μπούμε στην ουσία να ελέγξουμε τι ισχύει και τι είναι γεγονός και τι δεν ισχύει. Τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα και είναι χωριστή η εξουσία από την εκτελεστική. Μακάρι να συνέβαιναν έτσι τα πράγματα και στα δικά μας κρατη Εγώ πήγα στην Κολομβία με πολλές αμφιβολίες και επέστρεψα πεπισμένος ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναστείλουμε τη συμφωνία με την Κολομβία. Συναντήσαμε εκπροσώπους των, του Συνδικάτου Κότε που δεν είναι εκπρόσωποι των συνδικάτων, είναι εκπρόσωποι κομματικών και ιδεολογικών γραμμών. Και μας λένε όχι, μην υπογράψετε τη συμφωνία, γιατί τι θα κερδίσουν οι εργαζόμενοι. Όταν λοιπόν κάποιο αναφέρεται σε μια χώρα, θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση της χώρας αυτής. Είναι παράδοξο. Ε, που δεν επικρίνεται η Βενεζουέλα, για παράδειγμα. Μα η Βενεζουέλα ζει δικτατορία. Είναι χούντα ο Τσάβε στη Βενεζουέλα. Κανείς δεν το λέει αυτό. Πουθενά δεν γράφεται. Εγώ σήμερα μίλησα με τον Τζον Μόγκ και θα ήθελα να δω και άλλους συνδικαλιστές και δεν υπάρχει κανένας λόγος να επικρίνουμε συνεχώς εδώ πέρα την Κολομβία. Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από αυτή που περιγράφεται. Τώρα ο Ρίτσαρτ Χάουιτ θα συνοψίσει παρακαλώ. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους Επίτροπή και του συναδέλφου λίγο με απογοήτευσε ότι θα μου δώσατε λεπτομερεί απόψει ε, και θα ήταν ε, βοηθητικό αυτό για τη δουλειά μου αν είχαμε πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις έγκαιρα για σήμερα. Ίσως να μην περιμένετε οι δικές μας νομοδοτήσεις να είναι τόσο λεπτομερείς στις συστάσεις τους. Θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε τότε. Και λαμβάνοντας αυτό υπόψη θα ήθελα να σας καλέσω όχι απλά να στείλετε περαιτέρω σχόλια γραπτός, αλλά να έρθετε και να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εγκαίρως πριν από αυτή την προθεσμία που έχουμε για την υποβολή τροπολογιών. Και στον κύριο Μωράς που νομίζω από την ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου πραγματικά ε, με ανησυχεί το πώς εσείς ερμηνεύετε την παράγραφο 7. Είναι ήδη αρκετά δύσκολο σε αυτή τη μεγάλη ήπειρό μας να καταλάβουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Τώρα, αν οι δικοί μας συνάδελφοι ε, ε της Κομισιόν δεν διαβάζουν το κείμενο, τι να πω. Εδώ λέτε ότι εμείς συζητάμε δεσμευτικές στάνταρ, ενώ εδώ λέμε για εθελοντική προσπάθεια. Ε, στη δική σας συμβολή λέτε ότι η Κομισιόν θέλει να ενθαρρύνει ε, την τήρηση των εθελοντικών ε, προδιαγραφών. Εγώ λέω promote, προωθήσει. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είπατε και αυτό που είπα εγώ. Πραγματικά απογοητεύομαι. Ε, εγώ προσπαθώ να είμαι συμβιβαστικός όπου υπήρχαν προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τον Τζο Higgins που επικρίνει την Κομισιόν, νομίζω είναι αυτονόητα τα όσα ήδη είπαν μόνοι τους. Και θα ήθελα συγκεκριμένα και συμφωνώ μαζί του ότι είναι δίκαιο να πούμε πως έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα εντός της Ένωσης όσον αφορά το σεβασμό της, ε, των εθνικών προδιαγραφών εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων. Αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το επιβάλλουμε και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ελπίζω λοιπόν πως και άλλοι στην Επιτροπή θα το υποστηρίξουν, να μην επαναλάβουμε ένα λάθος όσον αφορά τις εμπορικές μας συμφωνίες. Ένα πρόβλημα δηλαδή που είχαμε εντός των δικών μας συνόρων. Και τώρα για το θέμα της Κολομβίας θέλω να χαμογελάσω σε σχέση με τα όσα είπε ο συνάδελφος ε, Φέμπρ. Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτά που είπε ή στις λεπτομέρειες που ανέφερε ο Χίγκινς εκείνος για το θέμα αυτό, γιατί εγώ κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτή η γνωμοδότηση και αυτή η έκθεση δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο εδώ για να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ πολύ σημαντικό θέμα και εγώ έχω πολύ έντονα συναισθήματα για την υπόθεση αυτή. και έχω διαμαρτυρηθεί κατά των των 2.700 θανάτων που δεν έχουν επιληθεί. Ε, όλα αυτά τα έχουμε καταγγείλει. Διάφορες ε, νομοθεσίες στην Κολομβία δεν είναι συμβατές με τις συμβάσεις ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Έχουμε διάφορες καταδίκες ε, σε σχέση με τις δολοφονίες και ο Ρίτσαρτ σωστά το είπε ότι δεν θα έπρεπε να, ε, να συμφωνήσουμε για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορία. Είναι όμως τεράστιο το θέμα. Δεν μπορούμε αυτό να το περάσουμε μέσω της εμπορικής μας πολιτικής και το πώς ε, θα ασχοληθούμε με τους συνδικαλιστές, τα υπόλοιπα κοινωνικά δικαιώματα. Ότι δεν πρέπει δηλαδή να το αντιμετωπίσουμε από την πίσω πόρτα. Δεν νομίζω πως αυτή η γνωμοδότηση είναι η κατάλληλη φάση για να πω ότι απλώς αναφερόμαστε σε κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την ε, αξιολόγηση βιωσιμότητας ε, που φαντάζομαι πως συμφωνείς μαζί μου και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση και έπειτα την ψηφοφορία για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Υπάρχουν τρεις υποθέσεις της Λιθουανίας, αλλά μόνο μία εντάσσεται εδώ σε σχέση με την, ε, τον κλάδο της κατασκευής κτηρίων. Θέλουμε να συμφωνήσουμε με αυτή την επιστολή εκτός από την παράγραφο 5. Αυτό που προτείνω λοιπόν να κάνουμε είναι εφόσον υπάρχει συμφωνία για το υπόλοιπο της επιστολής να ψηφίσουμε για την τροπολογία στην, στην παράγραφο 5 πρώτα και στη συνέχεια να ψηφίσουμε για ολόκληρη την επιστολή. Νόμιζα πως αυτό είχατε συμφωνήσει μεταξύ σας οι συντονιστές και έχει νόημα. Ναι, μισό λεπτό θα σας δώσω το λόγο παράγραφος 5 είναι η μόνη που, από ό,τι κατάλαβα έχετε πρόβλημα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αν υπάρχουν άλλες παράγραφοι εκτός από την 5 για την οποία έχετε πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Τσαμπαόρη χωρίς μικρόφωνο προς το παρόν. Ah, okay. Uh, Ευχαριστώ. Τώρα, ε, λοιπόν, δεν είναι εύκολη η θέση μου, διότι θα θέλαμε όλοι να φύγουμε νωρίτερα. Αλλά κοιτάξτε, κυρία Πρόεδρε, είναι θέμα αρχής αυτό. Βάζουμε μια ώρα για την ψηφοφορία και μια ημερομηνία και την ανακοινώνουμε και δεν την αλλάζουμε. Γιατί τώρα υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν άλλε υποχρεώσει την ίδια στιγμή και θα έρθουν στη συνεδρίασή μα όταν έχει προβλεφθεί η ψηφοφορία. Δεν είναι σωστό αυτό κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ να ε, σημειώσετε την απογοήτευσή μου, τη δυσφορία μου, τουλάχιστον να γραφτεί στα πρακτικά. Αυτό που εσεί οφείλετε να κάνετε ε, είναι ορθό, είναι να διατηρείτε και το χρονοδιάγραμμα και την ώρα και την ημερομηνία. αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία μας. Δεν μπορούμε κατά το δοκούν έτσι να αλλάζουμε και ψηφίζουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Όχι. Έχουμε προβλέψει μια ώρα για την ψηφοφορία. Η κυρία Γκρέσλε, για παράδειγμα, είναι σε εξωτερική ε, διοργάνωση, εκδήλωση του Κοινοβουλίου και θα έρθει την ώρα που είχαμε προβλέψει για την ψηφοφορία. Και τότε εμεί θα έχουμε πάει ήδη σπίτι μας. Παρακαλώ γραφτεί στα πρακτικά η έντονη διαμαρτυρία μου. Ναι. Το κατανοώ αυτό. Ε, όταν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να το σεβόμαστε. Αλλά ρώτησα τους άλλους συντονιστές και η πλειονότητά τους συμφωνούν να προταχθεί η ώρα της ψηφοφορίας. Το σημειώνουμε αυτό ότι έχετε αντιρρήσεις. Πριν από μια μισή ώρα περίπου ανακοίνωσα ότι ειδοποιήστε τις πολιτικές ομάδες γιατί θα ψηφίσουμε νωρίτερα και τότε κανείς δεν αντέδρασε. Και θεώρησα ότι είχαν όλη την ευκαιρία και ίσες ευκαιρίες να μαζέψουν τον κόσμο τους. Εάν κάποιοι είναι σε άλλες επιτροπές, είναι υποχρέωσή τους να, να έρχονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών και να είναι διαθέσιμοι την ώρα που συνεδριάζει η Επιτροπή. Ε, δεν το αλλάξαμε και πάρα πολύ, δεν, προτάξαμε πάρα πολύ την ψηφοφορία χρονικά. Ε, οι άλλοι οι συντονιστές συμφωνούν και παρακαλώ να προχωρήσουμε αν δεν έχετε άλλα σχόλια. Ο κύριος Σόρη, κυρία Πρόεδρε. Για τα πρακτικά το λέω. Κοιτάξτε, εγώ είμαι συντονιστή και εμένα δεν με ρώτησε κανένα ο συντονιστή. Επαναλαμβάνω, είμαι συντονιστή και δεν με ρωτήσατε. Μα η γραμματεία μου λέγει ότι δεν ισχύει αυτό. Ε, ε, ρωτήθηκαν οι συντονιστέ. και αν ήταν απόντες, ε, οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων είχαν ενημερωθεί ότι θα ψηφίσουμε νωρίτερα. Και ε, από τα όσα μου λέει η γραμματεία γνώριζαν όλες οι πολιτικές ομάδες το θέμα αυτό. Τώρα μου λέτε ότι δεν το γνωρίζατε. Το ανακοίνωσα επανειλημμένος, προηγουμένως, εδώ από το Προεδρείο και ε, ξέρω ότι οι περισσότεροι ήταν ενήμεροι ότι θα ψηφίσουμε νωρίτερα. Και είχαν οι πάλι της ομάδας σας την ευκαιρία να σας ενημερώσουν και να καλέσετε και τα μέλη σας να είναι παρόντα. Όταν κάποιος είναι μέλος σε μια επιτροπή, κανονικά φροντίζει να είναι και κοντά και να έρχεται. Ποιος θέλει τώρα το λόγο? Ο κύριος Τσάμπουνοκ. Κύριε eh, děkuji za slovo. Eh, vážená paní předsedající, Κυρία Πρόεδρε, Δεν έχω αντίρρηση να γίνει η ψηφοφορία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά ούτε και με μένα ήρθε κανείς σε επαφή, κανείς δεν ζήτησε τη γνώμη μου. Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Γενικά πάντως δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να θέτουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτή είναι η μία πιθανότητα. Ε, από την άλλη βέβαια θα πρέπει οι βουλευτές να είναι παρόντες ε, κατά τις συζητήσεις ε, της Επιτροπής μας. Όταν λοιπόν θέτουμε συγκεκριμένα χρονική στιγμή, τότε θα πρέπει να το τηρούμε. Ε, πρόεδρος, ε, σύμφωνα με τη γραμματεία, αν ε, δεν ρωτηθήκατε, είναι επειδή δεν ήσασταν παρόν και οι υπάλληλοι της ομάδας σας πρέπει να ενημερώθηκαν και είχατε μία μισή ώρα για να προσαρμοστείτε στο νέο χρονοδιάγραμμα. Έγινε η ανακοίνωση και εάν δεν ήσασταν εσείς παρόντε, θα έπρεπε οι υπάλληλοι τη ομάδα σα να επικοινωνήσουν μαζί σα και να σα ενημερώσουν. Ίσως θα πρέπει να συζητήσετε κάποια πράγματα με του υπαλλήλου τη ομάδα. Σα Πάντω η ανακοίνωση έγινε εγκαίρω. Ο κύριος Όρη. Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Ε, εντάξει, οφείλω να αναγνωρίσω ότι καθυστέρησα λίγα λεπτά. Ο αναπληρωτής συντονιστή ήταν παρόν και ούτε εκείνον το ρώτησαν. Ε, κάποια σφάλμα έχει γίνει, κάποιο λάθος έχει γίνει στη δικασία πέρα από αυτό. Είναι θέμα αρχής. Δεν είναι σωστό να βάζουμε ώρα για την ψηφοφορία και να την αλλάζουμε στην πορεία. Εντάξει, σημειώνω την κατάσταση. Τι να κάνω, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το ξέρω ότι θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες, αλλά θα λείπουν πολύ από την ψηφοφορία και σας το λέω. Και η δυσφορία μου διατηρείται ακέραιη. Ευχαριστώ. Each political group, that is all. If any other political group... Εάν ε, θέλει το λόγο κάποια άλλη πολιτική ομάδα, παρακαλώ να σκόσετε τα χέρι σας. Ε, αλλά να θεωρήσω ότι αν μίλησε ο συντονιστή κάποια πολιτική ομάδα, εκπροσωπεί όλη την πολιτική ομάδα. Υπάρχει κάποιο συντονιστή άλλη πολιτική ομάδα που θέλει να πάρει τον λόγο, αλλιώ να προχωρήσουμε στι ψηφοφορίε. Κανεί άλλο. Φοβάμαι ότι ήδη έχει μιλήσει ο συντονιστή σα. Ε, μόνο οι συντονιστέ θα μιλήσουν. Ε, αλλιώ προχωράμε στην ψηφοφορία. Έχουμε λοιπόν τη συζήτηση. Πρώτα και κατόπιν ψηφοφορία. Όσον αφορά την επιστολή λοιπόν, Είχαμε ομάδα εργασία. Η μόνη παράγραφο για, για την οποία υπάρχουν διαφωνίε είναι η παράγραφο 5. Εγώ θα ήθελα να ψηφίσουμε την, την παράγραφο 5 ω τροπολογία και να ψηφίσουμε κατόπιν το σύνολο τη επιστολή. Κυρία Μωράν, θέλετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όντως, Είμαι στην ομάδα εργασίας αυτή και μεταβαίνω τακτικότατα στις συνεδριάσεις και πρέπει να σας πω ότι η παράγραφος 5 έφτασε εκ των υστέρων μετά τη λήξη της ε, συνεδρίασης. Διερωτώ με λοιπόν με ποιο τρόπο έχει παρισφρήσει αυτή η παράγραφος ενώ είχαμε συμφωνήσει για μια γενική διατύπωση της επιστολής. Και ε, δεν έχω καταλάβει πώς έχει εμφανιστεί αυτό. Για ποιο λόγο. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που λένε εδώ είναι να αλλάξουν το ποσοστό στη συγχρηματοδότηση των μέτρων ΦΕΜ, e αλλά αυτό δεν είχε συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Anybody else wish to on that? Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Συμφωνώ, η κυρία Χάρκιν, συμφωνώ με την προγραλή σας. Αν δεν είχαμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό και να λάβουμε σωστή απόφαση. Εγώ τώρα το είδα και με προβληματίζει κάτι καινούριο να μας παρουσιάσετε τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε. Αυτό αποτελεί πρόβλημα. Η κυρία Κορνέλισον. Ναι. Ε, και εγώ έχω το πρόβλημα ότι η επιστολή δεν συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα. Το τανίστηκα από το κύριο μπροστά μου, αλλά μήπως μπορεί η πρόεδρος να το διαβάσει. Ναι. Ε, Κύριε Σέρκας, ποια είναι η θέση σας? My mistake. Mr. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Ο κύριος Σέρκας. Εγώ έχω πρόβλημα. Δεν έχω ούτε την επιστολή, ούτε ξέρω την παράγραφο 5 που λέτε. The difficulty, I'm told, is that we won't have the η δυσκολία από ό,τι μου λένε είναι ότι δεν θα έχουμε χρόνο, διότι θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε λέγει, θα πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα την επιστολή, να σας διαβάσω τη νέα παράγραφο αν αυτό σας βοηθάει. Από ό,τι καταλαβαίνω, η ε, ομάδα μελέτης έχει συναντηθεί αρκετές φορές και η μόνη παράγραφος για την οποία υπάρχουν διαφωνίες είναι η παράγραφος 5. Εάν σας βοηθάει, μπορώ να διαβάσω την παράγραφο 5 και την προτινόμενη νέα διατύπωση. Όταν θα την έχω διαβάσει, εάν θέλετε να την σχολιάσετε και πάλι, να έχουμε μια σύντομη συζήτηση, αλλά μου λένε ότι εάν δεν ψηφίσουμε τώρα την επιστολή, δεν, έχουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε στο μέλλον. Θα τη διαβάσω λοιπόν. Εάν θέλετε ε, να πάρετε το λόγο, μπορούμε να έχουμε μία σύντομη συζήτηση. Η παράγραφος θα έχει ως εξής, ότι ε, δυσαρεστείτε που το Συμβούλιο δεν ήταν διατεθειμένο να δεχτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να ε, ενισχύσει την ε, συγχρηματοδότηση στο 75% για τα μέτρα EGF για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη σε εποχές κρίσης ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί το σύνολο του δυναμικού του EGF για τους εργαζομένους και να αναπτύξει το επίπεδο των, ε, των, εργαζομένων. Η κυρία Μορέν. Σας ευχαριστώ. Εάν συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, αφαιρούμε τελείως το νόημα της ομάδας εργασίας το οποίο, στην οποία ε, έχουμε εργαστεί. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε η κυρία Αρκή. Σε αυτή την ομάδα εργασίας είμαστε λίγοι που αντιπροσωπεύουμε τα διάφορα κόμματα. Ε, έχουμε αφοσιωθεί σε αυτή τη δουλειά, έχουμε δουλέψει πολύ σοβαρά και αυτή η τροπολογία εμφανίζεται τελευταία στιγμή εδώ πέρα χωρίς ε, καμία ιδιαίτερη ε, αναφορά, ε, υπογραφή και νομίζω πως ε, μας βάζετε ενώπιον τελεσμένου γεγονότος αντίθετα κιόλα από τη δουλειά που κάνουμε συνήθως αυτή την ομάδα εργασίας. Πραγματικά βλέπω να παραμελείτε και να υπονομεύεται πλήρως η δική μας αφοσίλωση και η δουλειά που κάνουμε για αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω σε σχέση με τα όσο είπε η Ελιζαμπέτ. Δεν είναι γεγονός αυτό ότι ξαφνικά ε, εμφανίστηκε κάτι ε, στην επιστολή. Δεν είναι μόνο αυτό. Ε, υπάρχει συμφωνία διοργανική μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Και αυτή η νέα παράγραφος 5 ζητάει κάτι που παραβιάζει τη συμφωνία. Δεν μπορεί να παραμείνει στο κείμενο. Uh, uh, Κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Αλλά δεν ξέφρασε κανεί αντιρρήσει, όπω μου λέει η Γραμματεία. Τώρα, αφού όλοι σα ανησυχείτε τόσο πολύ για μια νέα τέτοια παράγραφο, Αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι επειδή η Κομισιόν έστειλε έτσι μια απάντηση. Αλλά να προτείνω έναν απλό τρόπο να προχωρήσουμε, αφού δεν σα δυσαρεστεί. Και αφόσον πρέπει να περάσει η επιστολή, α ψηφίσουμε για την τροπολογία στην παράγραφο 5. Και αν αυτό καταψηφιστεί, θα τηρήσουμε την αρχική παράγραφο 5 και θα ψηφίσουμε για ολόκληρη την επιστολή. Αν διαμαρτύρεστε επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει, η γραμματεία με διαβεβαιώνει ότι έχει κυκλοφορήσει. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω τη δική σας ε, οργή. Ε, το καταλαβαίνω, έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά. Αλλά η δυσκολία που έχουμε τώρα είναι ότι πρέπει κάποια επιστολή να περάσει. Ευχαρίστω να ψηφίσουμε ολόκληρη την πρωτότυπη επιστολή. Και αν θέλετε να τροποποιήσετε την παράγραφο 5, εντάξει, πάντως κάτι πρέπει να περάσει. Μπορούμε λοιπόν οι συντονιστές να λάβουμε μια σύντομη απόφαση, γιατί εσείς θα έπρεπε να το αποφασίσετε αυτό. Αν πιστεύετε δηλαδή ότι η ιδέα μου να ψηφίσουμε για τη νέα παράγραφο 5 και έπειτα στη συνέχεια για την επιστολή, το, ε, θα αρχίσει ο κύριο Σέρκα, μετά ο κύριο Σόρη και μετά η κυρία Χάρκιν κτλ. Μάλιστα. Υποστηρίζω πλήρως την πρόταση αυτή, αλλά κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να ξεκαθαριστεί. Αν ε, ε, στάλθηκε με ταχυδρομείο και αν είχαν ευκαιρία και χρόνο οι πολιτικές ομάδες στη διάθεσή τους για να το εγκρίνουν, να το απορρίψουν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, το διαδικαστικό. Επί της ουσίας είμαι υπέρ του κειμένου και θα το υπερψηφίσω. Μου λέγει η γραμματεία ότι την Τετάρτη απεστάλλει. Δεν είναι στα ντοσιέ, λέει η κυρία Όμεν. Ναι, αλλά την Τετάρτη τα στείλαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ορίστε, κύριε Ωρή. Ναι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει αρχίσει να χάνει τη σοβαρότητά της. Όλοι γνωρίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ήταν λεγόμενη τυρκουάζ ομάδα, εξοκοινοβουλευτικές δραστηριότητες είχαμε. Και εμείς έχουμε και εκλογέ, ξέρετε. Ε, ε, έχουμε επαφές με τους ψηφοφόρους μας, είμαστε εκτός και ξαφνικά μας στέλνουν με τόσο μικρή προθεσμία τέτοιο έγγραφο. Ουσιαστικά δεν έχουμε τις ε, ε, προϋποθέσεις για να ψηφίσουμε με τα λόγου γνώσεως αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Η κυρία Όμεν. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Διαδικαστικό είναι. Ναι, ναι. Άρθρο 172. Εντάξει, Πρόεδρε εδώ και καιρό δεν είμαι πλήρως, πλήρες μέλος. Ε, έρχομαι όμως. Ε, αλλά αυτή η σύγχυση που δημιουργείται είναι τρομακτική. Πέντε και τέταρτο ήρθα. Έπρεπε να είμαι εδώ για το προηγούμενο κείμενο, για την προηγούμενη έκθεση. Μπορεί να το έχετε στείλει. Αν δεν είναι στο φάκελο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσουμε. Και Επικαλούμε λοιπόν το άρθρο 172 εδάφιο δεύτερο που ζητεί ε, αναβολή της συζήτησης και της απόφασης για το θέμα αυτό. Σας εξήγησα ότι δεν μπορούμε να το αναβάλουμε αυτό, τη συζήτηση και την ψηφοφορία της επιστολής. Είμαστε υποχρεωμένοι. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρξει γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης υπομορφή επιστολής. Δεν τίθεται αυτό το θέμα, δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Αυτό που σας ζητώ είναι και προτείνω να αποφασίσουν οι συντονιστές αν θα ψηφίσουμε την παράγραφο 5 ως τροπολογία και μετά την αρχική επιστολή. Ο κύριος Σέρκας θεωρεί ότι είναι σωστό και συμφωνεί. Ο κύριος Άρη δεν ξέρω τι λέτε τελικά, αν συμφωνείτε ή όχι, αν θα πρέπει να ψηφίσουμε την παράγραφο και μετά την επιστολή ολόκληρη. Η κυρία Μωρέ φαίνεται να συμφωνεί, η κυρία Χάρκιν τι λέει. Συμφωνώ με την πρότασή σας, κυρία Πρόεδρε. se domnívám, že bychom Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τσάμπρονοκ. Να ψηφίσουμε μόνο την επιστολή όπως βγήκε από την ομάδα εργασίας, χωρίς την προσθήκη. Ο κύριος Έρι Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κανείς, κανείς δεν θέλει να αναβάλει, να καθυστερήσει ή να καταργήσει την επιστολή μας. Αλλά να ψηφίσουμε χωρίς την παράγραφο 5 που ξαφνικά ξεφύτρωσε μέσα στην επιστολή η Πρόεδρος. Κοιτάξτε. Επειδή τόσο πολύ ανησυχείτε για αυτή την πέντε, για να μπορέσουμε να περάσουμε κάτι, αν συμφωνούν και οι άλλοι ε, συντονιστέ, να ψηφίσουμε επί της επιστολής. Να μην ψηφίσουμε για την επιπλέον παράγραφο 5 Παρότι έχει κυκλοφορήσει, παρότι πρέπει να είναι στους φακέλους σας, διότι μοιράστηκε και στις αρχές της συνεδρίασης από ό,τι μου λέει η γραμματεία, αλλά αυτή είναι η απόφασή σας, να ψηφίσουμε μόνο επί της επιστολής που συμφώνησε η ομάδα εργασίας και στο μέλλον. Αν η γραμματεία μου λέει πως κάτι έχει σταλεί θα το πιστεύω και αν εσείς το έχετε τώρα ε, μπροστά στο έδρανό σας ή όχι είναι δικό σας πρόβλημα. Λοιπόν, να έχετε, να ρίχνετε μια ματιά στα mail σας για να είμαστε βέβαιοι πως δεν θα ξαναβρεθούμε σε αυτή την κατάσταση όπου οι μεν λένε ότι δεν έλαβαν ένα mail το οποίο έχει σταλεί Λοιπόν, μία ψηφοφορία θα γίνει και αυτή θα είναι επί της, αποστολής. Ποιοι, ε, επί της επιστολής ποιοι είναι υπέρ. Anyone against? Κατά κανείς. Abstentions. Αποχές. 39 uh, in favor. 39 υπέρ, ένας κατά και καμιά αποχή. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε στο επόμενο σημείο που είναι η απαλλαγή 2008. Και εδώ πολύ σύντομα συζήτηση για όλα τα θέματα για τον προπολογισμό. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Α, δεν είναι εδώ. Κύριε Όρη, θέλετε εσείς να συνοψίσετε. Δεν νομίζω πως είναι ιδιαίτερα επίμαχο το θέμα. Ε, ε, ε, Πρόεδρε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα καθόλου να πρέπει να κάνω σχόλια πριν την ψηφοφορία. Δεν ήταν τυχαίο που είπα στην αρχή ότι δεν συμφωνώ με την αλλαγή του ωραρίου, γιατί ήξερα ότι η κυρία Γκρέσλε ε, ε και δεν θα φτάσει εγκαίρως και δεν φταίει εκείνη. Αφού την έχουμε καλέσει για τα δε ώρα, έχει κανονίσει τι δουλειέ, τη, τι να κάνουμε τώρα. Θα ψηφίσουμε με τι συνθήκε αυτέ που επικρατούν. Απουσία τη κυρία Γκρέσλε. Ακριβώ η κυρία Γκρέσλε διαπραγματεύτηκε με του συναδέλφου μέχρι την τελευταία στιγμή και Ορίστε, τώρα θα γίνει ψηφοφορία απουσία της. Στις 2 το απόγευμα έγινε η τελευταία συνεδρίαση, δεν ξέρω τι έχει μεσολαβήσει εκ τότε. Oh. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Νταρντέν. Εγώ να επαναλάβω εξ ονόματο τη ομάδα μα ότι η βούλησή μα είναι βεβαίω η ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ελέγχου και αυστηρότητα στη διαχείριση των ταμείων και των διαφόρων γραφείων ε, και υπηρεσιών για να αποφευχθούν ε, οι απάτε, όπω σίγουρα είναι και η επιθυμία τη κυρία Γκρέσλε. Ισορροπία όμω με την αποτελεσματικότητα τη διαδικασία. Και πιστεύουμε πω η γνωμοδότηση δεν πρέπει να έχει στοχοδότηση να καταδεικνύει τη μια ή την άλλη την, την, την τάδε ή δίνα χώρα ή την τάδε ή δίνα οργανισμό. Και αυτό και έχουμε καταθέσει διάφορες τροπολογίες ώστε να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση και να ενθαρρύνουμε τη δουλειά των επιτόπου φορέων και να να ενισχύσουμε τις απαντήσεις ε, σε σχέση με τη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την κυρία Γκρέσλο μετά την κατάθεση των τροπολογιών μας ε, και μετά από τις διάφορες επαφές που είχαμε μαζί τις υποστηρίζουμε ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες αλλά όχι όλες. Εν πάση περιπτώσει, αυτές που δεν προσθέτουν κάτι νέο σε σχέση με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και θα ήθελα επίσης να προτείνω την ε, απόσυρση της τροπολογίας τρία σε σχέση με την ψηφοφορία για την απαλλαγή για την Επιτροπή. Αυτά, κυρία Πρόεδρε. Anybody else Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Από ό,τι καταλαβαίνω και η κυρία Φιγερέντο την έχει υπογράψει. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν και τη δική της άδεια για να, να, αποσύρετε την ε, τροπολογία. Και λείπει. Ας ψηφίσουμε αν δεν υπάρχουν άλλες ε, παρατηρήσεις. Πρώτα ψηφίζουμε απαλλαγή για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε τμήμα 3 ε, Επιτροπή. Ε, παράγραφος 3, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονικό έλεγχο να κάνουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Εάν δεν έχετε την κάρτα σας, σας παρακαλώ να μου κάνετε νόημα για να ψηφίσουμε, για να μετρήσουμε την ψήφο σα Σε λήξη τη ψηφοφορίας. Δεκάξι υπέρ, 24 κατά. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. ηλεκτρονικό έλεγχο. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 26 κατά. Τροπολογία 4. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εάν δεν έχετε την κάρτα, σας παρακαλώ πείτε μας αν ψηφίζετε υπέρ ή κατά. Ευχαριστώ. 36 υπέρ, μία αποχή, καμία ψήφος κατά. Ε, συγχαρητήρια στην κυρία Γκρέσλε. Η δεύτερη ψηφοφορία ε, έχει να κάνει με την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για το οικονομικό έτος 2008. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο θα κάνουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 3. Λήξη της ψηφοφορίας. Δεκαεννέα, δεκαεννέα, απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικό έλεγχο θα κάνουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 15 κατά. Χωρίς αποχές. 5, 6, 7 καταπίπτουν. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9-10 καταπίπτουν. 11 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο θα κάνουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 20-21. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Α, ζητώ συγγνώμη, δεν ψηφίζουμε την 12, πρόκειται για γλωσσική τροποποίηση. Λήξη, ε, συγγνώμη, ε, τελική ψηφοφορία για το σχέδιο χρωμοδότησης. Αρχή της ψηφοφορίας, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 13 κατά. Συγχαρητήρια και πάλι. Και πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2008. Ένα διαδικαστικό, η Ούμεν Ρόιτεν. Ναι. Ψηφίσαμε ένα σχέδιο που εγώ δεν έχω κάνει τις τροπολογίες του στο φάκελό μου. Τι γίνεται τώρα. Με ενημερώνουν οι τροπολογίε ήταν στου φάκελου σας. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Ομέν, εγώ στο δικό μου φάκελο δεν τι έχω τώρα. Mm. Ναι, μπορεί να μην τις έχετε, μες τις βάλαμε όμω. Λοιπόν, προχωρούμε. Ε, Πρόεδρε, η κυρία Ομέν, ψήφι υπέρ. Πρόεδρε, μια στιγμή, Πρόεδρε, ζητώ το λόγο. Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, λέγω. Μα είμαστε στη μέση μιας ψηφοφορίας. Ναι, αλλά απάντηση δεν πήρα. Μα το βάλαμε στο φάκελό σας. Ε, δεν είναι μέσα στο φάκελο. Τώρα τι θα γίνει. Έφερε τη στη μοναδική που δεν το πήρατε. Όχι, δεν είμαι η μοναδική. Εδώ, από αυτή την πλευρά της αιθούσης και σε διάφορες γλώσσες δεν έχουν την τροπολογία, τη τροπολογία στο φάκελο. Τώρα τις παίρνετε λοιπόν. Είναι επειδή ήρθατε καθυστερημένοι τις είχαν μοιράσει πριν φτάσετε. Πριν από μισή ώρα καταφτάσατε μόλις. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 1, αφού πήρε και η κυρία Όμεν Ρόιτεν τις ε, τροπολογίες. Καλό θα ήταν να έρχεται και νωρί και να τις παίρνει εγκαίρως. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχο θα κάνουμε. Vote Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται, λέει η πρόεδρος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ηλεκτρονικό έλεγχο θα κάνουμε για την τροπολογία 2. Αρχή της ψηφοφορίας. Συγγνώμη. Ευτυχώς που ελέγξαμε. 22 υπέρ. 20 κατά. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Η τέσσερα καταπίπτει και η τρία καταπίπτει. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 40 υπέρ. Μία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια και πάλι. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία 1. Αρχή της ψηφοφορίας. 25 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. Η 1, 2, 3 καταπίπτουν. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6 καταπίπτει και η 5 καταπίπτει. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι και η τελική ψηφοφορία μας έχει να κάνει με απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008. Η, στην πρώτη τροπολογία θα κάνουμε ξεχωριστή ε, ψηφοφορία Ξεκινάμε δηλαδή από το Notes the Course Findings, το σημειώνει τα αποτελέσματα του, του δικαστηρίου μέχρι την ε, ε, χρηστή οικονομική διακυβέρνηση στο μέλλον. Υπέρ του πρώτου μέρους, ε, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ του δεύτερου μέρους, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 39 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκρέσλε για την πολλή δουλειά που έχει κάνει. Συγχαρητήρια σε όλους σας.